Ας αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Θυμίζω, για σεβασμό των προσώπων, ότι η συνεδρίαση μεταδίδεται μέσω του ίντερνετ. με το έχετε Έχουμε τον πρόεδρο Φελίππο Γκοντζάλες μαζί μας σήμερα. Ένα έχει βέβαια. Ο άνθρωπο, αν ήθελε να διαβάσω όλου 10 λεπτά θα μου χρειαζόταν. απλώ. Σα θυμίζω τότε ότι στη διάρκεια τη προεδρία, του, τη Ισπανική Προεδρίας, τότε η Ισπανία μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό για μα, του ευρωβουλευτέ, είναι ο πιο σημαντικό τίτλο. σα είπα έχει πάρα πολλού τίτλου. προεδρεύει σε πολλά διεθνή όργανα κλπ. Αυτό είναι όμω το πιο σημαντικό. Πριν του δώσω το λόγο, είμαι υποχρεωμένος να τηρήσω την ημερήσια διάταξη. Και σας θυμίζω ότι το, έχει μοιραστεί το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης ήδη από τις 16 Σεπτεμβρίου. Ε, Σεπτεμβρίου. Έχουμε το χρονοδιάγραμμα για το 2011, προηγουμένως όμως καλύτερα να γίνουν οι συνεδρίες των συντονισμών. Σημείο 2, ανακοινώσεις, γιατί θεωρώ εγκεκριμένη την ημερήσια διάταξη. Το 2 λοιπόν Μία ανακοίνωση μόνο έχω. Από κοινού με τον πρόεδρο Αγγιλάρ στις 13 Ιουλίου γράψα μία επιστολή προς τον πρόεδρο Σαστέλ του Συμβουλίου και ζητήσαμε να μας δοθεί η εντολή του Συμβουλίου για την διαπραγμάτευση ένταξης της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη για την Προστασία των Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Η απάντηση που πήραμε στις 29 Ιουλίου με επιστολή, μάλλον μας ανακοινώθηκε άτυπα και με φύλαξη το περιεχόμενο αυτής της εντολής, ξαναγράψαμε επιστολή στις 29 Ιουλίου, οι δυο μας, προς το Συμβούλιο, θυμίζω συμβάλλει βάσει τη συνθήκη της Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να έχει κάθε πληροφόρηση πλήρη για τις πράξεις της Κομισιόν. Απάντηση πήραμε με επιστολή που πήραμε στις 30 Σεπτεμβρίου, όπου ο πρόεδρος της Επιτροπής των Μονίμων Αντιπροσώπων αναγνωρίζει εκ μέρους του Συμβουλίου το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να πληροφορείται άμεσα, αλλά διευκρινίζει ότι το έγγραφο μέχρι στιγμής ε, είναι εμπιστευτικό. Άρα μπορεί να δοθεί μόνο στους συντονιστές της Επιτροπής μας μόνο αφού υπάρχει μια αίθουσα στην οποία θα υπάρχει ειδική ασφάλεια να μην μπορούν να διαρρεύσουν πληροφορίες προς τα έξω μας λέει το Συμβούλιο θα μας δοθούν και άλλες πληροφορίες αναφέρεται στην Επιτροπή από το Συμβούλιο αλλά προφορικά σε συνάντηση με την Κομισιόν και, και κλεισμένων των θυρών. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να το μελετήσουμε το θέμα, όχι σήμερα βέβαια, όχι αυτή τη στιγμή. Στη συνάντηση με τους συντονιστές θα το θίξουμε. Τρία, τα πρακτικά έχουν μοιραστεί. Αν δεν υπάρξει αντίρρηση θα θεωρηθούν εγκεκριμένα. Και θα δώσουμε τώρα το λόγο στον πρόεδρο Φελίπε Γκοντζάλες. Σας θυμίζω όμως ότι η συνεδρίασή μας είναι ανοιχτή και σε πολλά μέλη άλλων επιτροπών για θέματα εξωτερικών, διεθνή θέματα, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Βιομηχανίας, Προσωρινή Επιτροπή για την Κρίση, Ειδική Επιτροπή για τις πολιτικές της Ένωσης μετά το 2013 Ήδη χαιρέτησα και προσωπικά και εκ μέρους σας τον πρόεδρο Φελίπε Γκοντζάλες. Ήρθε η στιγμή να του δώσουμε το λόγο. Ήδη γνωρίζετε ότι ο πρόεδρος Γκοντζάλες είναι επικεφαλής της ομάδας εργασίας που συνέστησε τον Δεκέμβριο του 2007 το Συμβούλιο για να μελετήσει την κατάσταση της Ευρώπης μετά το 2020. 2020-2030. Μπορεί η επιλογή και ο τίτλος να φαίνεται πολύ φουτουριστικός. Στην πραγματικότητα όμως, αυτά που συζητάμε σήμερα, οικονομικά, κοινωνικά, κράτος δικαίου, δίκηση, ενέργεια, ασφάλεια, καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας που είναι σημερινά προβλήματα που πρέπει να τα βλέπουμε σε μακρόπνοη προοπτική. Γιατί η πολιτική πρέπει να μπορεί να παρεμβαίνει όχι μόνο θεσμικά αλλά και μέσω σαφών ιδεών, μέσω προβλέψεων μεγάλου χρονικού βεληνικού. Ήδη συναντήσαμε τον πρόεδρο Γκονζάλε. Εγώ δεν είμαι πρόεδρο τη Επιτροπή μα βέβαια, αλλά είχε γίνει ήδη μια συνάντηση στι 21 Ιανουαρίου του 2009 για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Το ψήφισμα, το κείμενο παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο τη Ευρώπη στι 8 Μαου και τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα. Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε Γκονζάλε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε Κασίνη. Δεν ε, θα σας εξηγήσω ποιο είναι το περιεχόμενο της έκθεσης. Εξάλλου το έχετε στη διάθεσή σας από τον Μάιο. Μπορείτε να το διαβάσετε με την ησυχία σας. Όμως μπαίνω στον πειρασμό να δώσω μια εντύπωση ε, απεσιόδοξη για την Ευρώπη. Εγώ θέλω αυτή εξ αρχή να σας προειδοποιήσω ότι είμαι πεπισμένος για το ότι ζούμε σε μια υπερεθνική περιοχή με τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Την μεγαλύτερη ευημερία, την μεγαλύτερη ελευθερία. Έχουμε πετύχει δηλαδή υπέροχα πράγματα εδώ στην Ευρώπη. Καταφέραμε ε, από 12 χρόνες που είμαστε πριν από 20 χρόνια να γίνουμε 27 χώρες. Να έχουμε μια σταθερότητα στην Ευρώπη. Είμαστε σε μια ιστορική στιγμή που κανείς δεν φανταζόταν πριν από μερικά χρόνια. Και ακόμα και από τις Ηνωμένε Πολιτείε λένε ότι για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Ευρώπη δεν είναι ένα πρόβλημα, δεν είναι κάτι που ανησυχεί την Αμερική. Και μιλώ φυσικά για την Ευρώπη στο σύνολό της. Συγχρόνως όμως θα προσθέσω ότι ναι, ναι μεν δεν είναι πρόβλημα η Ευρώπη, αν εξαιρέσουμε βέβαια τα προβλήματα συντονισμού όσον αφορά την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, αλλά έλεγα δεν είναι πρόβλημα πια η Ευρώπη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά μέρος της λύσης. Αυτό λένε. Και κατά τη γνώμη μου, και εδώ έρχομαι να μιλήσω για τη δικιά μου τη δουλειά, ότι αρχίζουμε να χάνουμε λιγάκι την ε, σχέση μας με την παγκόσμια πραγματικότητα ή και με τον ίδιο τον πολίτη. Γιατί πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα όπως έχουν. Και τι μας λένε αυτά. Μας λένε ότι οι πολίτες δεν είναι τόσο πεπισμένοι υπέρ της Ευρώπης όπως ήταν πριν από 15 χρόνια. Και ότι σε διεθνές επίπεδο το ειδικό μας βάρος το οποίο δεν μετριέται από τον αριθμό των φωτογραφιών στις οποίες εμφανιζόμαστε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από τη δυνατότητα που έχουμε να επηρεάσουμε, να συναποφασίσουμε τις διάφορες διαδικασίες που οδηγούν στη νέα παγκόσμια πραγματικότητα. Εκεί είναι που νομίζω ότι χάνουμε λίγο έδαφος. Και άρα κάτι πρέπει να κάνουμε, να αντιδράσουμε. Σας παρακαλώ λοιπόν την ε, παρέμβασή μου εδώ, να μην την ερμηνεύσετε, γιατί θα μπορούσε κανείς να την ερμηνεύσει σαν απεσιόδοξη. Μην την ερμηνεύσετε έτσι, ότι της λείπει η αισιοδοξία. Όχι. Αλλά να τη δείτε σαν μια παρουσίαση που έρχεται από κάποιον που τον απασχολεί το μέλλον της Ευρώπης. Μιλάμε για τον ορίζοντα 2020-2030. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μιλήσουμε για το τι θα γίνει στην Ευρώπη το 2020-2030, αλλά πώς θα πάμε από τη σημερινή κατάσταση στο 2020-2030. Όταν ανέλαβα τη δουλειά αυτή, το είπα ήδη και το 2009, όταν ανέλαβα λοιπόν αυτή τη δουλειά, το Δεκέμβριο του 2007 που είχαμε την κρίση με τις υποθήκες κλπ. Έλεγα ότι είμαστε μέσα σε μια διεθνή οικονομική κρίση και δημοσιονομική, πρώτα δημοσιονομική, που δεν είχαμε ποτέ ζήσει, αλλά εξακολουθούμε να ζούμε. Επίσης είχα την αίσθηση ότι η συνθήκη της Λισαβόνας, που μόλις την είχαμε υπογράψει, την παραμονή, θα περνούσε από μια δύσκολη περίοδο επικυρώσεων και άρα από τη στιγμή που αφοσίζεται να δημιουργηθεί η ομάδα προβληματισμού και τη στιγμή που ξεκινάει να λειτουργεί η ομάδα αυτή προβληματισμού, ξέρετε ότι περνάει πολύ καιρό. Το, το Δεκέμβριο του 2008 αποφασίστηκε. Όμως, από τη στιγμή που αποφασίστηκε να φτιαχτεί μέχρι τη στιγμή που άρχισε να λειτουργεί η ομάδα αυτή, δεν είχαμε μόνο τις τοξικές υποθήκε, είχαμε και την κρίση της Lehman Brothers και είχαμε και την διεθνή οικονομική κρίση. Και πάλι το Δεκέμβριο του 2008 ε, πιστεύαμε, σε ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης τουλάχιστον, ότι το πρόβλημα ήταν βασικά πρόβλημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Όμω είναι προφανέ ότι όταν ξεκίνησε να δουλεύει η ομάδα προβληματισμού, καταλάβαμε ότι η οικονομική κρίση ήταν μεταδοτική, συστημική και παγκόσμια, αλλά ήταν μεταδοτική και έφτασε και στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν ήταν αδύνατον η ομάδα προβληματισμού να μην λάβει υπόψη τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης προκειμένου να καθορίσει τη στρατηγική της. Εξάλλου μέσα στην ομάδα υπήρχαν ορισμένοι ότι μα μην ασχοληθούμε με την κρίση γιατί σε 10 χρόνια θα φαίνεται γελίο να έχουμε συμπεριλάβει εμείς σε μια τέτοια έκθεση για το 2020-30 πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κρίση. Έτσι λέγανε ορισμένοι, αλλά δεν συμφωνούσαμε και εγώ δεν συμφωνούσα και φαίνεται αυτό σήμερα ότι δίκιο είχα. Διότι για την κρίση θα μιλήσουμε και φέτος και του χρόνου και σε 10 χρόνια και σε 20 χρόνια θα μιλάμε ακόμα για την κρίση και το 2029. Δηλαδή έναν αιώνα μετά, ε, από εκείνη την προηγούμενη κρίση του 2029, συνέχεια θα μιλάμε για την οικονομική αυτή κρίση. Η έκθεση βασίζεται και στην ιστορία. Για πρώτη φορά βλέπουμε ξεκάθαρα, εφόσον δεν το είχαμε προβλέψει αρκετά, ότι η κρίση καθορίζει τη νέα παγκόσμια πραγματικότητα. Δηλαδή, ποιες θα είναι οι καινούργιες τάσεις που θα αντιμετωπίσουμε. Προς τα πού θα κατευθυνθούν αυτοί που κερδίζουν και πού θα κατευθυνθούν αυτοί που χάνουν. Όλοι λοιπόν μιλάνε πολύ σοβαρά για αυτό το θέμα και λένε ότι το ειδικό βάρος περνάει από την Ευρώπη, τη Δυτική Ευρώπη, προς την Ασία προς τις αναδυόμενες χώρες οικονομικά. Και όλοι συμφωνούν ότι για το 70% της ανάπτυξης του ΑΕΠ ε, του παγκοσμίου τα επόμενα 15 χρόνια θα οφείλεται στις αναδυόμενες οικονομίες. Κανείς δεν αμφιβάλλει σήμερα για το ότι η Ιαπωνία, η οποία πριν από 20 χρόνια, 20 χρόνια μας φαινόταν ότι θα κατακτήσει την αγορά ολόκληρου του κόσμου, είναι τα 16 τελευταία χρόνια σε κρίση μέσα σε μια κρίση ή που δεν καταφέρνει να βγει ή που δεν θέλει να βγει από αυτήν. Κοιτάγαμε τι κάνει η Ιαπωνία και τα ίδια που λέγαμε πριν από 20 χρόνια για την Ιαπωνία τώρα τα λέμε για την Κίνα. Ότι η Κίνα θα τα σαρώσει όλα και θα είναι παντού. Το ίδιο λέγαμε και για τους Ιάπωνες πριν από 20 χρόνια. Ό,τι λέμε σήμερα για την Ιαπωνία θα λέμε σε 20 χρόνια και για την Κίνα, δεν το ξέρω. Πάντω η Ιαπωνία δεν φαίνεται να βγαίνει από την κρίση. Και οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρώπη μπήκανε σε κρίση. Και θα ήθελα να αναρωτηθούμε εμεί ω ε, Ευρωπαίοι, και το λέω και στην έκθεση, γιατί η Ευρώπη ω περιφέρεια, με διαφορέ που υπάρχουν μεταξύ των χωρών βέβαια, γιατί λοιπόν η Ευρώπη ε, αναλογικά πλήτεται περισσότερο και ζει πιο έντονα την οικονομική κρίση από ότι οι ίδιες οι Ηνωμένε Πολιτείε από όπου ξεκίνησε η οικονομική κρίση, η Λατινική Αμερική, η Ασία, που είναι και αυτές κάποιες περιφέρειες. Γιατί έχουμε την Ασιατική Βδομάδα εδώ στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, γιατί και ακριβώς επειδή δεν έχουμε την ε, απάντηση αυτή, ε, βλέπουμε τον κόσμο να χάνει την εμπιστοσύνη του κάπως. Πρέπει λοιπόν να καθίσουμε και να δούμε τι γίνεται στα διάφορα σημεία του κόσμου. Στην Ασία δεν πιστεύουν ότι τους έχει πλήξει η κρίση, πιστεύουν ότι ζουν καλύτερα από ποτέ και ότι το μέλλον είναι δικό τους. Στη Λατινική Αμερική, στη Βραζιλία για παράδειγμα, το ίδιο πιστεύουν. Και στην Ευρώπη, αυτό το οποίο διαπιστώνω εγώ και διαπιστώνουν όλοι, ανεξάρτητα αν λέμε τα πράγματα περισσότερο ή λιγότερο ομά, ε, περισσότερο ή λιγότερο απότομα, αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι οι Ευρωπαίοι της γενιάς μου, αλλά και της επόμενης, δεν λέω μόνο των νέων και τη επόμενη, πιστεύουν ότι τα παιδιά τους δεν θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες που είχαν ε, οι γονείς τους. Αυτή η κατάσταση επικρατεί στον κόσμο. Το αντίθετο δηλαδή από ό,τι συμβαίνει στην Ασία ή στη Λατινική Αμερική. Και το πώς αισθανόμαστε εμείς έχει να κάνει βέβαια με την πραγματικότητα που ζούμε. Ζούμε όμως όπως σας είπα καλύτερα από ό,τι ζουν άλλοι σε άλλα μέρη του κόσμου, αλλά έχουμε πολλές αφιβολίες για το κατά πόσο είμαστε σε θέση να διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο ζωής που έχουμε σήμερα. Το ίδιο παραγωγικό σύστημα που είχαμε μέχρι τώρα, το σύστημά μας κοινωνικής συνοχής Έχουμε αμφιβολίες, αμφιβολίες που είναι βάσιμες. Και εμείς στην ομάδα μας προσπαθήσαμε να δούμε πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι τόσο μια συζήτηση που θέλουμε να προκαλέσουμε. Θέλω όμως να ακούσω τη γνώμη σας. Γιατί δεν χρειάζεται να έρθω εγώ και να σας διαβάσω την έκθεση. Τη διαβάζετε μόνοι σας. 15 τέφχη είναι η έκθεση αυτή. Με διάφορα νούμερα. Για να δείξουμε ότι είναι όντως έτσι. Προσπαθήσαμε να καταδείξουμε το πρόβλημα και από εκεί και πέρα να συζητήσουμε και πάνω απ' όλα να πάρουμε αποφάσεις. Και πιστέψτε με, τα έχω πει και στο Συμβούλιο πριν από λίγο και στον Πρόεδρο του Συμβουλίου. Έχω κάνει και άλλες παρουσιάσεις σε διάφορους. Ε, λοιπόν, πιο πολύ απ' όλα με ενθουσιάζει η ιδέα του να έρθω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να παρουσιάσω τα συμπεράσματα της ομάδας μας. Γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να δημιουργήσει τον χώρο που χρειάζεται για να γίνει συζήτηση ευρεία με την κοινωνία των πολιτών και σε απλή γλώσσα. Στον καθένα να μιλάμε στη γλώσσα του. Γιατί προχωρήσαμε στη στρατηγική της Λισαβόνας χωρίς να πούμε στους πολίτες ότι είχαμε μια αποτυχία. Τώρα λοιπόν πρέπει να είμαστε ειλικρινεί και η πρότασή μας για το 2000-2010 να προχωρήσει έτσι ώστε να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες μας. Γιατί μην ξεχνάτε το 2000 για τη στρατηγική της Λισαβόνας είχαμε πει ότι θα γίνουμε η πιο μεγάλη δύναμη οικονομική που να βασίζεται στη γνώση. Ε, δεν γίναμε. Τι φταίει, η διάγνωση. Όχι τόσο. Εν μέρη. Είχαμε 29 στόχους. Δεν ήταν σωστή μέθοδος. Η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού, που σημαίνει ότι κάθε χώρα τελικά κάνει ό,τι της αρέσει, αν αυτό το συγκρίνουμε με τους 29 στόχους, αυτό τελικά σημαίνει ότι ο καθένας κάνει όντω ό,τι θέλει και από τα 29 σημεία σε τρία μόνο προχωρήσαμε. Σε σχέση με το 2000 δηλαδή, το σύνολο της Ένωσης δεν κέρδισε πόντους όσον αφορά τη θέση μας ως οικονομική δύναμη που βασίζεται στη γνώση. Όχι. Είμαστε ανάμεσα στην Αμερική και την Ασία. Και μας πιέζει η Ασία, η οποία προδεύει πολύ. Αυτή είναι μια κριτική, πρέπει να την πούμε στους πολίτες. Η στρατηγική της Λισαβόνας λοιπόν δεν δούλεψε. Και πιστεύουμε ότι δεν δούλεψε γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό. Η νέα λοιπόν στρατηγική τώρα, 2010-2020 της Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λιγότερου στόχου, γίνεται καλύτερο προσδιαρισμός. Ε, λοιπόν, αυτή η νέα στρατηγική θα είναι πιο αξιόπιστη. Γιατί παραδεχόμαστε ότι πριν δεν τα καταφέραμε. Τώρα, υπάρχει κάτι που με απασχολεί και το λέω σε όλους. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε σήμερα την κρίση και θα σας πω με ποια τρία στοιχεία και να καταπολεμήσουμε την κρίση η οποία είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Δεν είναι αλήθεια ότι την έχουμε αφήσει πίσω. Όχι, είναι εδώ μαζί μας σήμερα και θα είναι μαζί μας και στο μέλλον. Να φροντίσουμε για τις διαρθρωτικές αλλαγές εκείνες που έπρεπε να είχαμε κάνει πριν από 10 χρόνια, που πρόβλεπε η στρατηγική της Λισαβόνας και δεν κάναμε, έχουν μείνει πίσω. Και να αλλάξουμε και τη μεθοδολογία για την εφαρμογή της στρατηγικής. Δεν μπορεί να είναι ο ανοιχτό συντονισμό. Πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα με κίνητρα, για να μην πω με κυρώσει, ώστε να πάρουμε όλοι στα σοβαρά τους στόχους. Λέμε ανθρώπινο δυναμικό κλπ. κλπ. Ναι, αν δεν το κάνουμε, ή αν κάποιες χώρες, οι μισές χώρες δεν το κάνουν, τι θα γίνει, ε, τίποτα δεν θα γίνει. Και αν δεν γίνει τίποτα, η Ευρώπη με μια ενιαία νομισματική πολιτική και μέσα σε μια εσωτερική αγορά χωρίς ε, σύνορα θα χάσει οικονομικό συντονισμό, θα χάσει σε οικονομική αρμονία, άρα θα μείνει πίσω απέναντι στις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει. Όσον αφορά την κρίση, εγώ πιστεύω και είναι ένα από τα πράγματα που υπάρχουν ε, στην έκθεση και που μας διαφοροποιεί κάπως, δεν πιστεύω ότι πρέπει να σταματήσουν οι αντικυκλικές ε, πολιτικές μέχρι να έχουμε ανάπτυξη. Όμως αποφασίσαμε να σταματήσουμε τις αντικυκλικές πολιτικές. Αυτό είναι το τελευταίο. Και μας ήρθε από τον Ομπάμα, όχι, όχι, μη σταματήσετε τα αντικυκλικά μέτρα, διότι η παραγωγική οικονομία, η πραγματική οικονομία έτσι θα προχωρήσει. Ναι, και αυτό είναι το τελευταίο που θα σας πω. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι χώρες έχουν ένα περιθώριο ελιγμών για να κάνουν αντικυκλική πολιτική. Όχι. Γιατί? Γιατί όπως η δικιά μου χώρα τα δύο τελευταία χρόνια έχασαν το περιθώριο ελιγμών. Ήτανε ο καλύτερος μαθητής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και καταλήξαμε σε μια κατάσταση που δεν μας επιτρέπει να έχουμε περιθώριο ελιγμών για την αντικυκλική πολιτική. Κάποιες χώρες της Ευρώπης μπορούν. Αλλά κυρίως πρέπει να υπάρχουν ευρωπαϊκά μέσα. Και το λέω αυτό σε εσά τους ευρωβουλευτές να το σκεφτείτε και να δείτε τι θα κάνετε. Όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτά τα λέει η έκθεσή μας μέσα. Άρα λοιπόν... Μην γινόμαστε όμοιροι ορισμένων χωρών που έχουν χάσει το περιθώριο ελιγμών, υπάρχουν άλλες που δεν το έχουν χάσει και που θα μπορούσαν για ένα διάστημα να βοηθήσουν με τα αντικυκλικά μέτρα. Κάτι ακόμα. Κάνετε κάτι που αποκλίνει από αυτό που έχει αποφασιστεί. Τότε προσοχή, διότι δεν πρόκειται να έχουμε άλλη ευκαιρία. Θα έχουμε σαν τους Ιάπωνες ανάπτυξη. Δηλαδή μια μεσαία κατάσταση έτσι σημειωτών θα προχωράμε. Σύμφωνα με το πακέτο που προτείνουμε, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν είναι το υπεύθυνο για την κατάσταση που δημιουργήθηκε στην Ευρώπη με το ευρώ. Επιπλέον, το Σύμφωνο Σταθερότητας είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει νομισματική πολιτική. Αυτό όμως που φάνηκε από την κρίση είναι ότι δεν φτάνει. Συνεπώς, προτείναμε και γίνονται πράγματα. Προτείνουμε λοιπόν στην έκθεσή μας ότι πρέπει να προσθέσουμε στην νομισματική πολιτική και την νομισματική ένωση πολιτικές οικονομικής διακυβέρνησης για να μην αποκλίνουν οι πολιτικές μας. Υπήρχε μέχρι τώρα μια σύγχυση σε όλους μας, γιατί εμείς νομίζουμε ότι το πιο σοβαρό που συμβαίνει στην Ευρώπη, και έρχομαι στη δικιά μου τη χώρα, είναι η ανισορροπία των εθνικών δημοσιονομικών. Όχι, δεν είναι αυτό που μας οδήγησε στην κρίση. Αυτό που μας οδήγησε στην κρίση είναι ε, μία ανισορροπία ε, ισολογισμών 11-12%. Οι αποκλήσει στην οικονομία. Όχι η τήρηση, όχι του συμφώνου σταθερότητας που το 2007 στην Ισπανία είχαμε 2,5% παραπάνω ο ΑΕΠ και 37,5% χρέος σε σχέση με το ΕΠ. 4% ανάπτυξη και 5% ανάπτυξη της απασχόλησης. Πού να βρει κανείς καλύτερα στοιχεία από αυτά. Συγχρόνως είχαμε μια οικονομία, ένα εμπορικό έλλειμμα 10% και 11% στο ισοζύγιο πληρωμών. Συγχρόνως θα μπορούμε να κρατήσουμε μια νομισματική Ευρώπη σταθερή με αποκλίσεις τόσο μεγάλες στην οικονομική πολιτική. Συνεπώς η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται οικονομική διακυβέρνηση για την αγορά, για νομισματικούς λόγους κλπ. Γίνονται βήματα προς αυτή την κατεύθυνση σήμερα. Αλλά υπάρχει και ένα ερωτηματικό. Πρέπει να τροποποιήσουμε τις συνθήκες εγώ θα έλεγα καλύτερα να αφήσουμε ίσχυες τις συνθήκες για κάποιο διάστημα. Μην τις πειράξουμε. Διότι αν οι ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων αποφασίσουν και παρουσιάσουν μια οικονομική διακυβέρνηση και το Κοινοβούλιο συναποφασίσει με τους ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων, την έχουμε την ε, δυνατότητα στη συνθήκη της Λισαβόνας να προχωρήσουμε σε οικονομική διακυβέρνηση. Επαναλαμβάνω, να αρχίσουμε να πειράζουμε τη συνθήκη που κάποιος δεν θα επικυρώσει και κάποιος θα καθυστερήσει και δημοψήφισμα με δημοψήφισμα και δεν συμμαζεύεται, ας αφήσουμε τις συνθήκες την ησυχία τους. Θα μπούμε αλλιώ σε νέα κρίση. Δεν πειράζουμε τις συνθήκες. Και τέλος από το μέτρο, από τα μέτρα του πακέτου. Ε, μεταρρύθμιση στο δημοσιονομικό σύστημα. Η κρίση είναι η συνέπεια κακής λειτουργίας του συνολικού δημοσιονομικού συστήματος. Δεν έχουμε εναλλακτικέ. Τελείωσε αυτό. Οι ελάχιστες που υπήρχαν ήταν μια ουτοπία. Όμως δεν μπορούμε να καθίσουμε έτσι όπως είμαστε. Χρειαζόμαστε μια μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού συστήματος ώστε να αποφύγουμε εκ νέου να καταρρεύσει το σύστημα αν δεν υπάρξει μεταρρύθμιση, σε 7-8 χρόνια ετοιμάζεται, ψήνεται. Θα το έχουμε το επόμενο πρόβλημα. Οι τράπεζες, οι δημοσιονομικοί οργανισμοί βασίζονται σε εθνικούς κανόνες. Έτσι λειτουργούν, που διαφέρουν από χώρα σε χώρα του ευρώ. Δεν λέω της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικά, από τις χώρες του ευρώ μέσα. Η Ευρώπη λοιπόν θα έπρεπε να έχει μια μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού συστήματος που με μία φωνή έτσι ώστε όλοι να λένε τα ίδια να πηγαίνει η Ευρώπη στους G20 να συζητάει με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Οι Ηνωμένε Πολιτείες το ζητάνε. Οι αναδυόμενες χώρες δεν αισθάνονται καλά γιατί δεν είναι εκείνες που προκάλεσαν την κρίση. Και πιστέψτε με, περιμένουν η Βραζιλία και άλλοι που συμμετέχουν στους G20, περιμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη να προτείνουν κάτι λογικό το οποίο να επιτρέψει μια καλή λειτουργία του δημοσιονομικού συστήματος. Περιμένουν δηλαδή να προτείνουμε εμείς μια, ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα μας βοηθήσει να αποφύγουμε μια νέα κρίση, η οποία ετοιμάζεται σας λέω, ακολάπτεται. Στην επόμενη κρίση οι πολίτες δεν πρόκειται να ανεχτούν από μας να προσπαθήσουμε να σώσουμε τις τράπεζες όπως έγινε αναπόφευκτα αυτή τη φορά για να σώσουμε τις τράπεζες από τα δικά τους λάθη. Όχι, δεν θα το δεχτούν αυτό άλλη φορά. Μετά η έκθεσή μας περνάει σε κάτι που είναι πολύ γνωστό. Το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά, όλοι στην Ευρώπη. Τίποτα από αυτά που θα σας πω, είτε είναι η στρατηγική της Λισαβόνας, είτε η στρατηγική της Κομισιόν, ότι χρειάζονται διαφορετικές αλλαγές. Είναι γνωστό, ναι. Πρέπει να γίνουν γρήγορα και σε βάθος στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, στην Βόρεια Ευρώπη, κάτι έγινε. Καλό. Και γιατί. Γιατί εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε το δικό μας οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο. Είναι ένα μοντέλο που θέλουμε μιας κοινωνικής οικονομίας που να σέβεται το περιβάλλον. Για να πετύχουμε λοιπόν κάτι τέτοιο, πρέπει να έχουμε μία οικονομία πολύ ανταγωνιστική μέσα στην παγκοσμιοποίηση που ζούμε. Ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Και εφόσον δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί με χαμηλούς μισθούς, πρέπει να ανταγωνιστούμε με μεγάλη παραγωγικότητα με ποιότητα σε ανθρώπινο δυναμικό και με ε, τεχνολογίες εχμής. Αξίζει τον κόπο καυγάζει για αυτό το κοινωνικό-οικονομικό μοντέλο που το θέλουμε από παλιά και που μας οδήγησε στην ευημερία και την κοινωνική συνοχή που έχουμε σήμερα. Ναι, αλλά δεν μπορεί να είναι το ίδιο τον 21ο αιώνα, γιατί τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οπότε η ιδέα πρέπει να είναι αυτή. Για να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι η οικονομία έχει γίνει μια οικονομία καζίνο χωρίς κανόνες, προσπαθώντας να αντισταθμίσουμε τις ανισορροπίες που δημιουργήθηκαν σε όλα τα συστήματα. Με την παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε αυτό. Φροντίσαμε να υπάρχει μεγάλη διευκόλυνση δανεισμού με πολύ χαμηλό κόστος. Ο κόσμος λοιπόν δεν βελτίωσε τις δικές του δυνατότητες στην πραγματικότητα, αλλά αύξησε τις δυνατότητες του δανεισμού, χρέωσης του. Αυτό έκανε. Αυτό είναι το μοντέλο. Το οποίο οδήγησε την αναπτυγμένη Δυτική Ευρώπη και Δυτικό κόσμο σε μια κατάσταση που θα έχει να πληρώνει τις επόμενες δεκαετίες. Κίνα, μεγαλύτερη παραγωγός χώρα, που είναι και μεγαλύτερη, θα γίνει σε λίγο και η μεγαλύτερη χώρα ε, που καταναλώνει, θα έχει τη μεγαλύτερη κατανάλωση δηλαδή ως χώρα σε λίγο, θα γίνει και ο μεγαλύτερος πιστωτής σε λίγο στον κόσμο. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια κοινωνική συμφωνία την οποία θα φροντούσε να βάλει από την αιγίδα του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να βελτιωθεί η παραγωγικότητα, η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και έτσι να μπορέσουμε να τροποποιήσουμε το παραγωγικό μας μοντέλο. Βάσει αυτόν που πιστεύουμε. Και εδώ έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Στα 100 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου έχουμε λιγότερα από τα μισά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κέντρα αριστείας δεν έχουμε λοιπόν και πολλά. Αν αναρωτιόμασταν από αυτά τα φαινόμενα Google, Microsoft, πώς από αυτά είναι ευρωπαϊκά. Πώς στην Ευρώπη φτιάξαμε κάτι τέτοιο. Πού στην Ευρώπη. Amazon για παράδειγμα λοιπά δεν έχουμε πολιτιστικό τελικά χώρο μέσα στον οποίο να αναπτυχθούν τέτοιες δραστηριότητες. Αυτό είναι το τραγικό. Έτσι εμποδίζουμε πρωτοβουλίες οι οποίες μπορεί να είναι πολύ καλές και κρατάμε τις άχρηστες. Οι πέντε μεγάλες ε, επιχειρήσεις στην Ευρώπη που είχαμε πριν από 20 χρόνια, 30, είναι ίδιες και σήμερα. Δεν έχουν αλλάξει, ενώ στην Αμερική, στην Ασία έχουν αλλάξει. Υπάρχει καινούριο αίμα, με τεράστια επιτυχία. Έπειτα, βλέπω ότι συζητιέται σε όλες τις χώρες όποια και αν είναι η κυβέρνηση στην κάθε χώρα, τα πράγματα αλλάζουν και οι κυβερνήσει δεν αντιμετωπίζουν τα μεγάλα προβλήματα. Για παράδειγμα, τη γύρανση του πληθυσμού. Δουλεύουμε λιγότερο, ζούμε μέχρι τα 80. ...70 εκατομμύρια θα έχουμε στον, ε, λιγότερο θα έχουμε στον ενεργό πληθυσμό το 50. Και 90 εκατομμύρια περισσότερο κόσμο. Τα παιδιά δηλαδή που τώρα πάνε σχολείο, όταν θα φτάσουν να πάρουν σύνταξη, πάρα πολύ δύσκολα θα είναι τα πράγματα. Η αναλογία δηλαδή ανάμεσα στον ενεργό πληθυσμό και τον μη ενεργό θα είναι κάτι τρομερό. Πολύ ωραία που αυξάνει το προστόκιμο ζωής και η ποιότητα ζωής. Βεβαίως, πολύ θετικό το βρίσκω αλλά σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα αντιστάθμισμα. Η πυραμίδα δηλαδή αλλάζει σχήμα. Μπαίνει η κορυφή στη βάση και η βάση στην κορυφή. Χρειάζονται λοιπόν διάφορες πολιτικές, υπάρχει μέσα στην εκθεσή μας και διάφορα για τις γυναίκες, για τα παιδιά. Ωραία. Αλλά υπάρχει και κάποια σκέψη για τη μετανάστευση, τις μεταναστευτικές ροές. Τη σήμερον ημέρα, όποιος μαζεύει ψήφους, κάνει, ε, μιλάει κατά της μετανάστευσης. Δεν έχουμε λύση λοιπόν για το μεταναστευτικό παρά μόνο εάν φροντίσουμε να έχουμε μια σοβαρή μεταναστευτική πολιτική. Αυτά βέβαια δεν συζητιούνται σήμερα και θα έπρεπε να συζητιούνται. γιατί δεν είναι το 2025 που πρέπει να κάνουμε τις πολιτικές μας για τη γύραση του πληθυσμού και τη μετανάστευση. Τώρα πρέπει να τις κάνουμε αυτές. Το 2025 θα είναι πάρα πολύ αργά. Δεν θα έχει τίποτα να κάνουμε τότε. Σας είπα λοιπόν για το οικονομικό μοντέλο, για το ανθρώπινο δυναμικό, σας είπα για το δημογραφικό σύστημα. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα στην έκθεση. Τα πυρηνικά. Τι κάνουμε με την ενέργεια και τις κλιματικές αλλαγές. Θα αρχίσω από το τέλος. Η Ευρώπη έχει την πιο προηγμένη κοινή θέση όσον αφορά την καταπολέμηση των, κλιματικών, των κλιματικών αλλαγών. Σε σχέση με τον κόσμο ολόκληρο. Ε. Το Δεκέμβριο όμως στην Κοπεχάγη η Ευρώπη δεν μέτρησε. Μηδέν. Και θα σας πω ποιο είναι το μυστικό. Άλλο είναι να έχει καλή κοινή θέση και άλλο πολύ διαφορετικό είναι να έχεις μια κοινή στρατηγική για να υποστηρίξεις τα ευρωπαϊκά συμφέροντα απέναντι στους συνομιλητές σου. Και αυτό δεν το είχαμε. Ούτε ενεργειακή κοινή στρατηγική έχουμε, ούτε κοινή στρατηγική για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Έχουμε μια κοινή θέση και αυτό μας φτάνει. Και έπειτα πάμε στην Κοπεχάγη και εκεί όλα είναι ήδη έτοιμα. Η Κινέζοι τοποθετούνται, ο Ομπάμα που την έκανε. Οι τρεις λοιπόν μεγάλοι παίκτες λένε τι πρέπει να γίνει και εμείς πρέπει να το δεχτούμε ή να μην το δεχτούμε. Είναι το ενεργειακό σοβαρό, ναι. Ελπίζω ότι θα τηρήσουμε τους στόχους μας 2020 και το 2030 να είμαστε λίγο πιο φιλόδοξοι ακόμα. Πάντως το 2030, να ξέρετε, εκτός αν βέβαια γίνει μια τεχνολογική επιστημονική επανάσταση, που βέβαια δεν μπορεί κανείς να το προβλέψει. Αλλιώς λοιπόν το 2030 η παγκόσμια εξάρτηση από τα στερεά ορυκτά θα είναι 80%. Αν προχωρήσουμε όπως πάμε τώρα. Άρα λοιπόν η ενεργειακή πολιτική έχει τεράστια σημασία. Χρειάζεται λοιπόν αποταμίευση, χρειάζεται αποτελεσματικότητα. Αλλά πρέπει να διαπραγματευτούμε και με τους προμηθευτές μας. Η κάθε χώρα θέλει να κρατήσει τις δικές της δυνατότητες. Δεν γίνεται έτσι. Γιατί 80% των Ευρωπαίων πολιτών δεν ενισχύουν την ε, θέση της Ευρώπης. Έχουμε 15 εκατομμύρια καταναλωτές. Αλλιώς θα διαπραγματευτούμε με τους ε, Ρώσους όλοι μαζί από ότι κάθε μία χώρα μας χωριστά. Δεν το κάνουμε όμως. Αυτή είναι μια τεράστια ενεργειακή πρόκληση για την οποία κατά τη γνώμη μου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο. Να φροντίσει ώστε να τηρηθούν οι στόχοι 2020. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κέρδισε σε εξουσίες μετά την Λισαβόνα και εκπροσωπεί και τους ε, Ευρωπαίους πολίτες που ψηφίζουν ε, τους Ευρωβουλευτές. Άρα λοιπόν μπορεί να βοηθήσει σε αυτούς τους στόχους. Και υπάρχει και κάτι ακόμα. Αλλά πρώτα μία παρατήρηση για την εσωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας. Όταν μιλάμε για την εσωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, ακόμα και στην εντολή του Συμβουλίου, το μόνο που βρίσκουμε είναι την απειλή από την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα. Σίγουρα είναι η πιο ξεκάθαρη απειλή που έχουμε μπροστά μας. Αλλά οι άλλες ξαφανίστηκαν. Κρίση στη Γεωργία. Τίποτα. Δεν περιγράφω τώρα τίποτα. Το αναφέρω ότι υπάρχουν κι άλλα δηλαδή που θα έπρεπε να σημειώνονται. Στην έκθεση δεν είναι πολύ καθαρό, τέλος πάντων να βρούμε συνένεση μεταξύ 12. Τέλος πάντων, θα έπρεπε να έχουμε και μια πολιτική γυτνίασης, ιδιαίτερα δυναμική. Δεν μπορεί στις σχέσεις μας με τη Ρωσία να τις βλέπουμε τον ίδιο τρόπο όπως με την Νότια Αφρική, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανένα, η Νότια Αφρική φυσικά είναι αδειόμενη χώρα πολύ σημαντική. Αλλά με τη Ρωσία πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη σχέση. Άρα τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να αναπτύξουμε αυτή τη σχέση. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια στρατηγική για τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας, πολύ προσεκτική, γεμάτη περιεχόμενο. το ίδιο και με κάτι άλλο που είναι περισσότερο εσωτερική πολιτική παρά γετνίαση. Τι κάνουμε με την Τουρκία. Τι θα κάνουμε, θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο ή θα μείνουμε πιστοί στις δεσμεύσεις που πήραμε πριν από 10 χρόνια. Κάποιοι από τους ηγέτες που συμφώνησαν με τη συμφωνία τότε, τώρα τους βλέπω κατά. Εγώ έφυγα πριν από τον κόλ. Αλλά Αλλιώς είχαν τα πράγματα τότε. Τότε λέγαμε ότι η θέση της Ευρώπης δεν ήταν αρκετά όρημη ώστε να γίνει υποψήφια χώρα η Τουρκία. Όταν όμως αποφασίστηκε ότι είναι υποψήφια χώρα η Τουρκία, δεν μπορεί τώρα να αλλάζουμε. Πρέπει να είμαστε συνεπείς με αυτό που αποφασίσαμε. Και σας το λέω, αν είχε μείνει παραπάνω ο Κολ μπορεί να μην είχε συμφωνηθεί αυτό. Δεν ξέρω. Πάντως, κι εγώ ήμουνα αρκετό καιρό πρόεδρος. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε συνεπείς με τις αποφάσεις μας. Γιατί αυτό που γίνεται με την Τουρκία είναι πολύ πιο σοβαρό. Αυτό που γίνεται με την εξωτερική της πολιτική, με την ε, νέα της στάση στον κόσμο. Τη νέα θέση που αποκτάει στον κόσμο. Εμείς δεν βλέπουμε σε βάθος, δεν θέλουμε να ξέρουμε τίποτα. Έτσι, 20 χρόνια θα διαπραγματευόμαστε για να πούμε τελικά πως όχι. Θέλω να πω και κάτι που δεν το θίγουμε γιατί δεν θέλαμε να θίξουμε θεσμικά ζητήματα. Η Ευρώπη φτιάχνει την εξωτερική της υπηρεσία, υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αποφασίζει κανονικά, αλλά θα συναποφασίσει για την υπηρεσία αυτή, γιατί πρέπει να εγκρίνει τον προπολογισμό για αυτή την υπηρεσία. Συνεπώς, μέσα από τις αρμοδιότητες που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποφασίζει και για αυτή την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Ε, λοιπόν, με πονάει, αλλά πρέπει να σας πω ότι κάποιος πρέπει να είναι επικεφαλής. Δεν μπορεί, ξέρετε, σε ένα Υπουργείο Εξωτερικών ο Υπουργός διατάσσει. Στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης όμως βλέπω ότι έχουμε να κάνουμε με έναν αυτόνομο οργανισμό. Αυτόνομο σε σχέση με τι, για ποιο πράγμα. Αν θα κάνει την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, δεν μπορεί να είναι αυτόνομο. Ορίζουμε έναν ύπατο για να συντονίσει έναν αυτόνομο οργανισμό. Όχι. Αν ήταν για την εμπορική πολιτική, που είναι κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής μπορεί ή την πολιτική συνεργασίας που είναι μέρος της εξωτερικής πολιτικής αλλά που έχει τους αρμόδιους επίτροπους κάθε φορά. Αλλά μία είπατε εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική δεν ξέρω που θα καταλήξει αυτή η υπηρεσία εξωτερικής δράσης αλλά για μένα θα είναι ό,τι πιο αναποτελεσματικό μπορεί να υπάρξει. Έτσι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια κοινή εξωτερική πολιτική. Είπα πολλά, το ξέρω, αλλά αυτά ήταν μόνο τα κύρια στοιχεία. Για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν τόνοι εκθέσεων, τόνοι στοιχείων για τη μετανάστευση, για την εξέλιξη των εκπαιδευτικών μας συστημάτων, του ανθρώπινου δυναμικού, για την παραγωγικότητά μας, ανά άτομο, ανά ενεργό, ανά δεν ξέρω τι, για την ανταγωνιστικότητά μας στην παγκόσμια οικονομία, για την λειτουργία του κράτους ευημερία. Πληροφορίες έχουμε για τα πάντα. Αυτό που δεν έχουμε είναι συντονισμό από την Ευρώπη της πληροφορίας αυτής, ώστε να πάρει σάρκα και ώστα ως ένα σχέδιο. Ευχαριστώ πολύ. Μακάρι να τα καταφέρει η Ευρώπη. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε Γκονσάλες για την παρέμβασή σας και την δουλειά που έγινε πιο πριν, την ομάδα που συνέταξε το πρόγραμμα αυτό Ευρώπη 2030 που είναι ένα έγγραφο σύντομο σε σχέση με αυτό που μας εξηγήσατε, όπως μας εξηγήσατε σε σχέση με τις, τον όλο προβληματισμό. Η ομάδα σας Ευρώπη 2020-2030 έχει ένα προφητικό χαρακτήρα που συνδυάζεται βέβαια με εργαλεία. Να γίνουν οι προβλέψεις, μετά χρειάζονται όμως εργαλεία για να εφαρμοστεί η πολιτική. Μας αναφέρετε τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου στο μέλλον η Ευρώπη να είναι σύμφωνη με τα αρχικά οράματα των ιδρυτών της. Έχω αναφέρει ονόματα συναδέλφων που θα μιλήσουν πρώτος ο συνάδελφος Νταφ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς κύριε Κονσάλης για την ανάπτυξη του θέματος και την έκθεσή σας την οποία ανέγνωσα καθώς επίσης ευχαριστώ και για την κριτική που ασκείται στην παρούσα κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις γειτονικές της χώρες. Συμφωνώ πλήρως σχετικά με την στρατηγική σημασία της Τουρκίας. Λυπούμε δε που μέρος της εντολής σας σας απαγορεύει να μιλήσετε για θέματα συνόρων. Βέβαια γνωρίζουμε τους λόγους και δεν χρειάζεται να επανέλθω. Το υποβόσκον πρόβλημα των σχέσεων Τουρκίας-Ευρώπης εξακολουθεί να υπάρχει και μάλιστα η βαρύτητά του αυξάνει καθώς προχωρούμε στην προσπάθεια να στερεώσουμε τη θέση μας στην Ήπειρο. Σχετικά τώρα με την δημοτικότητα και νομιμότητα του Κοινοβουλίου του οποίου ενισχύθηκαν όντω οι αρμοδιότητες με την συνθήκη της Λισαβόνας. Έτσι λοιπόν η θεσμική του νομιμοποίηση είναι ασφαλής. Αλλά εξακολουθούμε να μην έχουμε την αξιοπιστία, την δημοτικότητα που θα θέλαμε στα μάτια του κοινού. Θα ήθελα να μάθω από εσάς. Τι σκέφτεται η ομάδα σας σχετικά με το θέμα αυτό. και ιδιαίτερα τι πιστεύετε για τον ρόλο των πολιτικών κομμάτων και την συγκριτική αδυναμία των ευρωπαϊκών ομοσπονδιών κομμάτων που έχουμε όπως το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το Κόμμα Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, Φιλελευθέρων κλπ. Θεωρείτε ότι μια ενδεχόμενη αλλαγή στην εκλογική διαδικασία μέσα από την οποία βγαίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις εκλογές του 2014 που να φτιάξει μία ε, πανευρωπαϊκή εκλογική περιφέρεια εκλέγοντας ορισμένους βουλευτές από μια υπερεθνική λίστα, από ένα υπερεθνικό ψηφοδέλτιο, θα μπορούσε να αποτελέσει θετική συμβολή στην βελτίωση της ε, νομιμοποίησης του Κοινοβουλίου. Της δημοτικότητας δηλαδή και νομιμοποίησης του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Ντάφ. Ε, η κυρία Γκουρμάη, Αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τα περισσότερα από όσα αναπτύξατε κύριε ε, Πρόεδρε Γκονζάλες. Πρόκειται για σημείο καμπής στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απαντήσεις που θα δοθούν στην κρίση πρέπει να συνδεθούν και με μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές θα είναι πιο δύσκολες από ό,τι θα ήταν για παράδειγμα στις ΗΠΑ η Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ετερογενής, αν και όλο και πιο ενωμένη πολιτικά. Είναι ένα πρακτικό παράδειγμα μια συνεργασίας. Κάτι το οποίο είναι καλό για μια χώρα δεν είναι απαραίτητα καλό για όλους μακροπρόθεσμα. Μιλώ για το εθνικό και το ευρωπαϊκό συμφέρον και την ενδεχόμενη βάση για μια συμφιλίωση. Όταν οι ιδρυτές πατέρες κατενόησαν ότι εκχωρώντας ένα μέρος της, μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα μπορούσαν να ασκήσουν ωστόσο οικονομική και πολιτική επιρροή που δεν θα είχαν διαφορετικά και ο λόγος της ε, πορείας Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακριβώς αυτός ότι βρέθηκε δηλαδή πάντοτε ένα συμβασμός. Γι' αυτό και είμαι πεπισμένη ότι στο τέλος η Ευρώπη θα μπορέσει να αναμορφώσει τις κοινωνίες της και την οικονομία της να ξαναπαίξει τον ηγετικό της ρόλο στον κόσμο. Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένας διαρκής επανακαθορισμός. Αλλά να πούμε ακριβώς ποια είναι τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Είναι όλων τα εθνικά συμφέροντα. Η έκθεσή σας είναι ένα σημείο αφετηρίας, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτά που ξεκινήσατε εσείς. Πώς το βλέπουν τα όργανα που εκπροσωπούν τις εθνικές κυβερνήσεις. Πώς θα ρίξουν το φως της συζήτησης. Εγώ είμαι μάλιστα και εισηγήτρια για την πρωτοβουλία των πολιτών που είναι νέο όργανο το οποίο προσφέρει η ε, συνθήκη της Λισαβόνας στους Ευρωπαίους πολίτες. Μιλήσατε και για αξίες. Περνούμε μια κρίση ευρωπαϊκών αξιών είναι αρνητική, αρνητικός αντίκτυπος του ανεξέλεγκτου νεοφιλελευθερισμού. Πώς μπορούμε να πείσουμε χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα ότι χρειάζεται μια οικονομική διακυβέρνηση, ρύθμιση δηλαδή των αγορών. Επίσης, πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε την διστακτικότητα των πολιτών. Για παράδειγμα, μόνο 42% πήγαν να ψηφίσουν στις τελευταίες ευρωεκλογές. Πιστεύω ότι η έκθεσή σας είναι ένα εξαιρετικό σημείο αφετηρίας. Και ένα μικρό σχόλιο. Εάν συγκρίνετε την στρατηγική τη Λισαβόνα και την ευρωπαϊκή στρατηγική του 2020, με ποιον τρόπο, βέβαια αυτή ε, ξεκίνησε ήδη από την Ισπανική Προεδρία. Πιθανώς ε, να έχουμε λιγότερες αξίες, όχι 29 αλλά μόνο 5, αλλά θα πρέπει να πείσουμε και το υπόλοιπο του πληθυσμού. Ευχαριστούμε την κυρία Γκουρμάη. Ε, Ευχαριστώ. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας εκ μέρου πολλών Ισπανών Ευρωβουλευτών ότι νιώθουμε περήφανοι που αναλάβατε εσεί επικεφαλή αυτής της ομάδας προβληματισμού και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε σήμερα μαζί μας. Σε αυτή τη συζήτηση για την Ευρώπη πρέπει να έχουμε πιο συχνά επαφές. Εποφελούμε από αυτή την ευκαιρία για να πω ότι αυτά που είπατε για τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον όλο προβληματισμό τα βρήκα πολύ ενδιαφέροντα. Όντω, η θήκη τη Λισαβόνα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ένα ρόλο και πρωτοβουλία και προώθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Γι' αυτό λοιπόν θέλω τέσσερα πράγματα να πω. Πρώτον, σε σχέση με τη διεύρυνση και όχι μόνο για την Τουρκία, εσείς πώς βλέπετε την διεύρυνση της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένων και των Βαλκανίων δηλαδή, η Κροατία σχεδόν σίγουρα θα μπει όπου να είναι. Με 30-32 χώρες πώς βλέπετε εσείς τη διευρεμένη Ευρώπη όταν ξέρουμε την εμπειρία που έχουμε με τις 27 χώρες μέλη. Μήπως η Ευρώπη έτσι πάει σε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων πιο πολύ. Σε διάφορους τομείς, τους οικονομικούς με την Ευρωζώνη πρώτα απ' όλα, αλλά και σε άλλους. Μήπως τελικά καταλήξουμε να έχουμε μια Ευρώπη με διαφορετικές ταχύτητες που να μην ε, έχει όλες τις χώρες να προχωράνε με τον ίδιο ρυθμό. Κάτι άλλο που δεν είπατε, αλλά υπάρχει στην έκθεσή σας, είναι τα δικαιώματα στην ηθαγένεια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε φτιάξει μια εσωτερική αγορά όπου κινούνται πάρα πολύ εύκολα τα εμπορεύματα, τα κεφάλαια, αλλά δυσκολευόμαστε πάρα πολύ για να αντιμετωπίσουμε και να αντισταθούμε στις... στα κράτη-μέλη, για να πετύχουμε την ε, ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Σε θέματα γάμων, σε θέματα κληρονομιά, σε θέματα αναγνώρισης πανεπιστημιακών διπλωμάτων, σε θέματα ε, αναγνώρισης ε, πτυχίων, επαγγελματικών προσόντων. Εκεί δεν έχουμε μια ενωμένη Ευρώπη. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να φροντίσουμε περισσότερο για την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Εκεί που τώρα πάμε τόσο αργά. Τρίτον, συχνά, και εγώ το έχω πει σε εσά, ότι εσείς λέτε ότι φτιάχνουμε τις βάσεις για τη νέα δημοσιονομική φούσκα. Πού? Πού αυτή τη στιγμή μπαίνουν οι βάσεις για μια νέα οικονομική κρίση. Πώς θα έπρεπε να αντιδράσει η Ευρώπη για να αντιμετωπιστεί αυτή η νέα φούσκα. Τέλος, η οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη σίγουρα είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε. Το Συμβούλιο φτιάχνει κάτι που το ονομάζει Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Σε αυτή την έννοια συμπεριλαμβάνουμε τις δημοσιονομικές προσεγγίσεις των κρατών μελών έτσι ώστε να τηρηθεί καλύτερα το σύμφωνο σταθερότητας. Μέσα σε αυτό το ευρωπαϊκό εξάμεινο, είναι η ερώτησή μου, θα φτιάξουμε τις διαρθρωτικές δομές ώστε να συμπεριλάβουμε τα κίνητρα ή τις κυρώσεις που δεν θέλετε να τις ονομάσετε κυρώσεις, ώστε τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν σε διαρθρωτικές αλλαγές. Και τέλος, νομίζετε ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια προεδρία του ΕΚΟΦΗΝ, μια δηλαδή οικονομική αρχή η οποία να έχει την ευθύνη διακυβέρνησης των 27 ε, ή μάλλον των 16 οικονομιών. Εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει μια τέτοια μορφή. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο σε άλλους συναδέλφους, θεωρώ σκόπιμο ο πρόεδρος Γκοζάλης να απαντήσει σε αυτές τις τρεις πρώτες παρεμβάσεις. Απαντήσει κατά ομάδα, κατά κάποιο τρόπο. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Πρώτον, για την Τουρκία, στην έκθεση τα λέμε ξεκάθαρα για να συμπληρωθεί η διαδικασία διαπραγματεύσεων και η προσχώρηση. Δεύτερον, το θέμα της νομιμότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο έχει νομιμότητα, αδιαφυσβήτητα, γιατί εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία. Έχει και θεσμική νομιμότητα στην άσκηση των ε, καθηκόντων του που προβλέπεται από το συνθήκη της Λισαβόνας. Αν του λείπει κάποια νομιμότητα, αυτή θα ήταν η νομιμότητα της δράσης. Και αυτή εξαρτάται από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι θα κάνει. Από την, τη δικιά μου πολιτική εμπειρία ξέρω ότι η πρώτη νομιμότητα είναι μια προϋπόθεση. Αλλά η νομιμότητα μέσω της δράσης είναι η ικανή. Υπάρχει ικανή και αναγκαία. Η μία είναι ικανή, η άλλη είναι αναγκαία. Μόνο εφόσον υπάρχουν και οι δύο, μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένο. Εμείς φροντίζουμε λοιπόν για αυτή τη νομιμότητα που να βασίζεται στη δράση. Δεν είμαι εγώ που θα απαντήσω. Οι ίδιοι ευρωβουλευτές είναι που πρέπει να απαντήσουν σε αυτό. Και έτσι φτάνω και στα πολιτικά κόμματα στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι θα ήταν καλό να υπήρχαν 30, 40 ή 50 ε, σε κάθε πολιτική ομάδα εκλεγμένοι από ολόκληρη την Ευρώπη. Και να είναι και υποψήφοι για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μην υπάρχει πια σύγχυση. Υπάρχει αυτή η εναλλακτική σοσιαλδημοκράτες, χριστιανοδημοκράτες, ε, συντηρητικοί κτλ. Δεν παρουσιάζω λοιπόν μόνο υποψήφιους και πρόγραμμα, αλλά συγχρόνως και κάποιον επικεφαλής που θεωρώ ότι θέλω να προεδρεύσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, η μεταρρύθμιση στην Ευρώπη είναι πιο δύσκολη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφίβολα. Η διαδικασία λήψη αποφάσεων στην Ευρώπη είναι κάτι πιο περίπλοκο. Ανέλησα κάπως και αναλύω την κρίση στην Καλιφόρνια. Ακούγεται ανέκδοτο, αλλά είναι αλήθεια. Που έχει το πιο ψηλό ΕΠ κατά κεφαλή στον κόσμο. Κι όμως, τα προβλήματά της δεν μπορεί να τα λύσει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Προϋπολογισμός για την εκπαίδευση είναι πιο κάτω από ό,τι για τις φυλακές. Είναι σε μια κατάσταση κρίσης χωρίς διέξοδο. Τα δύο τρίτα του Κοινοβουλίου εγκρίνουν τον προπολογισμό. Και η πρωτοβουλία πολιτών κόβει τον κανόνα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Φτάνουν δηλαδή στο Κοινοβούλιο διάφορες πρωτοβουλίες οι οποίες εγκρίνονται με πλειοψηφία και γίνονται νόμος χωρίς κανείς να ασχοληθεί με την οικονομική στήριξη του μέτρου, με τον προπολογισμό. Αυτά συμβαίνουν στην Καλιφόρνια, που είναι το πιο πλούσιο η πιο πλούσια πολιτεία των Ηνωμένων αλλά και στον κόσμο, αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει λύση στο σύστημα τους. Επιστήνω λοιπόν την προσοχή σας στο γεγονός ότι στη δικιά μας αντιπροσωπευτική δημοκρατία, που τόσο έχει προχωρήσει, αρχίζουμε να διακρίνουμε προβλήματα σοβαρά διακυβέρνησης. Και ορισμένοι όχι εγώ και προσοχή τι όρο χρησιμοποιούμε, ορισμένοι αρχίζουν να βλέπουν πολύ θετικά τις κινέζικες προοπτικές. Δεν είναι κάτι που θα αγνοήσουμε, θα αφήσουμε στην πάντα. Επανέρχομαι. Η εμπειρία που έχουμε από την Ευρώπη, που είναι ε, κυριαρχία ε, μοιρασμένη μεταξύ μας. Αυτό τουλάχιστον είναι το μεγαλύτερο ρεύμα. Έχει πρόβλημα όχι μόνο λήψης αποφάσεων, όχι γιατί το Συμβούλιο πολύ συχνά αναλύει τα προβλήματα τα οποία εξετάζουμε και είναι ξεκαθαρή στην ανάλυση τους. Άρα την κατανόηση και τον εντοπισμό του προβλήματος τα έχουμε, δεν είναι αυτά που με απασχολούν. Αυτό που με ανησυχεί εμένα είναι η βούληση. Μια φορά που έγινε γνωστό το πρόβλημα, που το καταλάβαμε και που έχουν ληφθεί αποφάσεις, εφαρμόζονται. Δεν είναι πρόβλημα εξυπνάδας να το βρήκαμε το πρόβλημα ή όχι, το βρήκαμε. Πώς θα εφαρμόσουμε τη λύση. Έχουμε τη θέληση να βρούμε τον προπολογισμό για παράδειγμα. Θα δείτε στην έκθεση ότι άπαξ και πάρθει κάποια απόφαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να φτάσουμε σε ένα ποσοστό επενδύσεων ως ένα από τα στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε ανταγωνιστικότητα κτλ. Αυτό δεν σημαίνει ότι στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε την υποχρέωση να καλύψουμε αυτό το στόχο. Αν όμως το Συμβούλιο Συμβούλιο είμαστε όλοι, γιατί είπαμε ότι είναι μοιρασμένη η κυριαρχία, έτσι. Ε, δεσμευτεί υπέρ ενός τέτοιου στόχου ή οποιοδήποτε άλλου, πρέπει να έχει στήριξη από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, αλλά και από τον προϋπολογισμό των 27 χωρών των οποίων οι επικεφαλείς δέχτηκαν ότι πρόκειται για προτεραιότητα. Άρα δεν φτάνω στο τελευταίο τμήμα, δεν ξέρω, στο, ευρωπαϊκό εξάμεινο ή κάποια άλλη στιγμή, προσοχή, μην μπερδεύουμε την οικονομική διακυβέρνηση με την ε, διακυβέρνηση του προπολογισμού. Πριν σας είπα ότι η οικονομική και δημοσιονομική διακυβέρνηση ε, πρέπει να βοηθάει να τηρείται το σύμφωνο σταθερότητας αλλά χρειάζεται σύγκληση των οικονομιών. Έτσι. Τώρα για το ευρωπαϊκό αυτό εξάμεινο που μου λέγατε. Αν ε, αναλάβουμε τη δέσμευση τα επόμενα χρόνια η κάθε κυβέρνηση θα λέει πρέπει να πετύχουμε τέτοιο ποσοστό δημοσίων επενδύσεων. Λέω για παράδειγμα έτσι. Πρέπει να υπάρχει όχι μόνο ο αντίστοιχος προπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος στο κάτω-κάτω θα είναι το 1% αντί για το 24-25% της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των Πολιτειών. Όχι, με αυτό το, 20, το 1% δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει καμία πολιτική. Η φιλοδοξία μετριέται με το χρήμα που βρίσκεται από πίσω. Η ομάδα μου δεν μπορούσε να προτείνει περισσότερα χρήματα για τον Ευρωπαϊκό Κορβανά, αλλά αυτό που σας λέω είναι ότι οι ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων που αναλαμβάνουν τη δέσμευση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για ένα συγκεκριμένο ποσοστό για δημόσια επενδύσει, για παράδειγμα, πρέπει αυτό να ανταποκρίνεται και στους εθνικούς προπολογισμού. Να αντικατοπτρίζεται και σε αυτού. Τώρα, αν είμαστε 30-32 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα αλλάξει βασικά το σημερινό μας πρόβλημα. Κάτι άλλο με απασχολεί. ανεξάρτητα από την Τουρκία. Όποια και αν είναι η καινούργια χώρα που θα μπει, φέρνει μαζί της ένα εθνικό πολιτιστικό ή εθνικό θρησκευτικό που μπορεί να δημιουργήσει αποκλεισμού. Πέρα από τη δυσκολία της Τουρκίας, βλέπουμε ότι τα Βαλκάνια μπαίνουν Έχουν όμως μαζί κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πολιτιστικά κλπ. Μιλήσατε για την Ευρώπη πολλών ταχυτήτων. Πάντα στην Ευρώπη είχαμε πολλές ταχύτητες στην διαδικασία της οικοδόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλες πολλές ταχύτητες, άλλες περιόδους πολλών ταχυτήτων είχαμε και το παραδεχόμασταν όλοι, άλλες υπήρχαν χωρίς να τις αναγνωρίζει κανείς. Συμβαίνουν αυτά. Και με τα δημοψηφίσματα που άλλο δεν κέρδιζαν, άλλο δεν κέρδιζαν. Οι opting out, άλλοι που βρίσκονται επικεφαλής του ΝΑΤΟ και όμως έχουν opting out. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η μεταβλητή έτσι κι αλλιώς. Και μπορούμε να διατηρήσουμε αυτή την κατάσταση υπό τον όρο ότι δεν θα είναι τόσο μεταβλητή ώστε να καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τελικά κανείς δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει ο ίδιος ή οι υπόλοιποι. Πρέπει να μπορούμε να διαχειριστούμε την ποικιλομορφία καταστάσεων. Διαφορετικές καταστάσεις θα υπάρχουν. Άλλοι είναι μέσα στο ευρώ, άλλοι δεν είναι μέσα στο ευρώ. Το ίδιο και για θέματα ασφάλειας. Υπάρχουν ουδέτερες χώρες διαφοροποίησεις υπάρχουν. Από όλα, ό,τι θέλετε υπάρχει εδώ μέσα. Τα πάντα. Υπάρχουν ε, λοιπόν πολλές και διαφορετικές καταστάσεις. Μπορούμε να οργανωθούμε με αυτές, ναι. Μπορούμε να αποφασίσουμε ότι οι διαφορές δεν θα είναι τόσο μεγάλες, ώστε η τελική διακυβέρνηση να γίνεται ουτοπία, να μην είναι εφικτή. Τώρα, έχουμε νομισματική ε, μονάδα. Έχουμε το Eurogroup με το ευρώ. Μερικές φορές σκεφτόμαστε, αφού υπάρχει πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να μας εκπροσωπεί, ο πρόεδρος ολόκληρου του Συμβουλίου θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι είναι και επικεφαλής της οικονομικής ζώνης του ευρώ αλλά και της άλλης. Δεν χρειάζεται να έχουμε χιλιάδες πρόσωπα. Τώρα, του ορίζουμε και μετά την επομένη τους λέμε «Α, όχι, εσύ υπάλληλο που σε κλέξαν οι υπόλοιποι». Αποδυναμώνουμε έτσι τα όργανα μας. Το βασικό είναι, και πρέπει να σας το πω, ότι τη μεγαλύτερη εξουσία την έχει αυτό εδώ το όργανο στο οποίο βρίσκομαι εγώ. αν θα υπάρχει καινούργια οικονομική κρίση. Το έχω πει ότι κολλάπτεται και δεν το λέω εγώ, το λένε πολλοί ειδικοί, στον τύπο θα το διαβάσετε. Και γιατί. Γιατί το μόνο που έχει αλλάξει από τη λειτουργία του δημοσιονομικού συστήματος που μας οδήγησε στην κρίση είναι ο περιορισμός των πιστώσεων υπέρ της παραγωγικής οικονομίας. Αυτό είναι το μόνο που έχει αλλάξει. Κατά τα άλλα τα προϊόντα, τα παράγωγα, τα χρηματοοικονομικά, τα swaps, ε, όλα αυτά, τρίχες. Οι επικεφαλής των τραπαζών, κάποια ηλικία και πάνω, το γνωρίζουν πολύ καλά, ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα, εξακολουθούν να πολλούνται. Εδώ η τράπεζες επενδύσεων μα οδήγησαν σε αυτή την κρίση. Και εμεί τα έχουμε βάλει με τη Lehman βρόμαν, Brothers. Όχι, όχι. Στην τράπεζα που ο πελάτης αποτελεί μόνο το όργανο για να πετύχει το προϊόν, είναι το πρόβλημα. Κανονικά έναν πελάτη με τις αποταμιεύσεις του πρέπει να τον συμβουλέψω τι να τα κάνει τα λεφτά του και στον άλλον θα δώσω ένα δάνειο φροντίζοντας να μην τον καταστρέψει η επιστροφή των χρημάτων. Έτσι θα έπρεπε. Έτσι θα έπρεπε να δουλεύουν οι τράπεζες. Αλλά τελικά τα προϊόντα, τα τραπεζικά διαλέγουν τον πελάτη και έχει τον άποδο. Και γιατί, γιατί υπάρχουν τα μπόνους. Δεν θα πάρει κανείς μπόνους αν ε, δεν ε, προχωρήσει το προϊόν που θέλει να προωθήσει. Και τελικά αγοράζουν οι πελάτες των τραπεζών οικονομικά προϊόντα που καλά καλά δεν ξέρουν τι είναι. Τώρα, είναι ιταλική ιδέα, η ιδέα της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, Είναι αλήθεια. Εφόσον, αν είχε πετύχει αυτό, δεν θα χρειαζόταν τίποτα άλλο. Η ιδέα είναι ταλική, λοιπόν. Προχώρησε λίγο. Θα μπορούσε να έχει προχωρήσει περισσότερο, ναι. Αλλά είναι δύσκολο να καταλάβουμε πώς είναι δυνατόν σε μια περίοδο που η τεχνολογία μας βοηθάει να προχωράει η πληροφορία σε χρόνο μηδέν, να μην έχουμε προχωρήσει στα κοινωνικά δικαιώματα μεταξύ όλων. Θα έπρεπε να υπάρχει δυνατότητα. Εφόσον ένα πολίτη σε μια χώρα έχει το ένα και το άλλο κοινωνικό δικαίωμα, αυτόματα θα πρέπει να το έχει και στην άλλη χώρα. Δυστυχώς δεν προχωρήσαμε σε αυτό. Και χειρότερα υπάρχουν και πιο γελία. Μιλάμε για την κινητικότητα μέσω του Εράσμους και άλλων προγραμμάτων. Όταν ένα ζευγάρι όμως, είτε άντρα γυναίκα, είτε άντρα άντρας, ε, Γάλλος, Πανός, πάνε στην Αγγλία. Κυκλοφορούν έτσι, μέσα στην Ευρώπη. Αν αποφασίσουν να φτιάξουν οικογένεια δεν ξέρουν ποιο είναι το δίκαιο το οποίο εφαρμόζεται στην περίπτωσή τους. Ποιο αστικό δίκαιο. Αν είμαστε από δύο διαφορετικές χώρες και ζούμε σε μια τρίτη χώρα, δεν ξέρουμε τι ισχύει για αυτούς. Θα έπρεπε να διευκολύνουμε τη ζωή των νέων που κυκλοφορούν μέσα στην ευρωπαϊκή επικράτεια που θέλουμε να την νιώθουν δικιά τους. Είναι ένα ανθρώπινο δράμα το οποίο μπορεί να λυθεί. Μόνο εμπόδια όμως υπάρχουν σήμερα και όχι λύσεις. Η εσωτερική αγορά είναι ένα τεράστιο πράγμα. Το νέο νόμισμα είναι επίση κάτι καταπληκτικό. Η ελευθερία διακίνηση πάρα πολύ καλά στην Ευρώπη. Όλα αυτά είναι επιτεύγματα. Και όλα αυτά τα φτιάξαμε, όχι από πάνω προ τα κάτω, όπω θα έλεγε και ο Σολάνα, πρέπει να ξεκινάμε το χτίσμα από κάτω προ τα πάνω. Μερικέ φορέ το ξεχνάμε πρέπει να πηγαίνουμε στον πολίτη και να του λέμε Εσύ που είσαι πολίτη, τι ανάγκε έχει. Όχι επιχειρηματία, όχι ο πάροχο υπηρεσιών, όχι δεν ξέρω εγώ ποιο. Να ξεκινάμε από κάτω. Ποιε είναι οι ανάγκε του πολίτη. Δεν το κάνουμε. Δεν θα έπρεπε να ρωτάμε τον πολίτη πρώτα ποιε είναι οι ανάγκε του και από εκεί να αρχίζουμε να φτιάχνουμε. Και είναι λογική. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Και εγώ ω πρόεδρο προσπαθώ αυτό να κάνω. Πρόεδρο προβληματισμού. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, ε, πέντε συνάδελφοι είναι γραμμένοι. Παρακαλώ να είστε σχετικά σύντομοι. Γιατί στι πέντε θα πρέπει να αρχίσουμε τις ψηφοφορία Γιάννης Μπερνοεύο πρώτος. Ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ τον Πρόεδρο Κονσάλες που ήρθε εδώ σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διάβασα την έκθεση το Μάιο, μάλιστα. Η πρώτη μου παρατήρηση είναι ότι υπέβαλε την έκθεση αυτή σε ένα συμβούλιο το οποίο ήταν περιγμένο από την οικονομική κρίση. Και σε ένα άρθρο στη χώρα μου διάβασα ότι το Συμβούλιο δεν θα έδινε και τόσο μεγάλη σημασία σε αυτό γιατί είχαμε την κρίση την ελληνική του ευρώ θα παίρναγε στα ψηλά. Ναι. Ο πρόεδρος Κονζάλες είναι επικεφαλής μια ομάδας προβληματισμού. Μπορεί να το ξέρει αυτό ο πολίτης. Σίγουρα δεν ξέρει όμως ότι έχει υποβάλει και έκθεση. Εγώ δεν ξέρω. Μπορεί να υπάρχει και να μην το ξέρω εγώ. Κάποια επίσημη απάντηση, αντίδραση από το Συμβούλιο το οποίο έθεσε σε εσά και στους σοφούς την εκπόνηση αυτής της έκθεσης ή από την Επιτροπή. Υπήρξε κάποια αντίδραση. Κάτι πρέπει να πούνε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ναι, ασχολήθηκε. Θα έπρεπε να ασχολείται περισσότερο και να δίνει περισσότερη προσοχή. Αλλά εσείς που ήσασταν ε, εδώ, το είπατε, ότι το Κοινοβούλιο έχει κερδίσει εξουσίες, ναι, αλλά θα θυμόσαστε πάρα πολύ καλά ότι το Συμβούλιο είναι εκείνο το οποίο κολλάει στα πράγματα και δεν προχωράει. Μερικές φορές ασχολούνται μόνο με την τιμή του μπακαλιάρου. Λέτε ότι κάνετε τη διάγνωση, αλλά συγχρόνως προτείνετε και λύσεις. Μεταρρύθμιση, είπατε προτείνει η έκθεσή σας. Πιο πέρα όμως, πώς μπορούμε να αντιδράσουμε στην εθνικοποίηση ή επαναθνικοποίηση των διαφόρων πολιτικών ή και στα μέτρα που παίρνουν διάφορες χώρες και ακούγονται στα μέσα ενημέρωσης όπου ακούσαμε πολιτικούς που λένε οι Βρυξέλλες με υποχρέωσαν. Λες και οι ίδιοι δεν συμμετείχαν στις συνεδριάσεις όπου ελάμβανταν αυτές ε, οι αποφάσεις, αλλά όταν τι εφαρμόζουν στις χώρες του και ο κόσμο διαμαρτύρεται, λένε Α, οι Βρυξέλλες με αναγκάζουν. Και είναι από όλο το πολιτικό φάσμα, έτσι. Δεν είναι μόνο ενό χρώματο. Πολλά σχόλια θα είχα να κάνω, αλλά τέλος πάντων. Ένα ακόμα. Για το θέμα της μετανάστευση, απασχόλησης, ανταγωνιστικότητας ενέργεια, κλιματικές αλλαγές Όλα αυτά που μας είπατε Μα είπατε ότι δεν θα τα λέγατε επειδή τα λέει η έκθεσή σα, αλλά τελικά η παρουσίασή σα ακολούθησε ακριβώ τον άξονα τη έκθεσή σα. Μια κάπω αισιόδοξη παρατήρηση. Εγώ έχω ασχοληθεί με τα εξωτερικά ζητήματα, ακόμα και σήμερα. Απ' έξω μας βλέπουν κάπως καλύτερα από ό,τι βλέπουμε εμείς από μέσα τα πράγματα. Είναι συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες λέτε λαμβάνονται πιο εύκολα οι αποφάσεις από ό,τι εδώ. Μα ίσως αποφάσεις που δεν είναι σε βάθος. Οι μεταρρυθμίσεις όμως του Ομπάμα ξέρετε πολύ καλά ότι είναι αντιμέτωπε και όχι μόνο αυτή για την υγεία αλλά και άλλες και μικρές μεταρρυθμίσεις είναι αντιμέτωπε με τεράστια εμπόδια στι Ηνωμένε Πολιτείε και υπάρχουν μεγάλε καθυστερήσει και στι Ηνωμένε Πολιτείε. Και εκεί είναι περίπλοκη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Και εκεί μιλάνε ορισμένοι για την παρακμή των ΗΠΑ. Τέλος για τις αναδυόμενες χώρες. Ξέροντας την ιστορία της οικονομίας και την εξέλιξη των χωρών μας, οι χώρες BRIC για παράδειγμα, δεν έχουν πάντα σχέση μεταξύ τους. Μερικά πράγματα ναι, Ινδία, Ρωσία, Κίνα. Τα επόμενα 20-30 χρόνια δεν θα περάσουν από μια σημαντική κρίση θα συνεχίσουν την ίδια ανάπτυξη που είχαν τα τελευταία 10 χρόνια, εγώ πιστεύω πως όχι. Ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με οικονομική κρίση και εκείνη. Αυτά είναι μερικέ σκέψεις που είχα να σας μεταφέρω και ευχαρίστω να ακούσω τα σχόλιά σα. Ευχαριστώ, ο κύριο Σέρκες, και ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο Γκονζάλες που ήρθε. Σύμφωνο με του συναδέρφους και εγώ σα ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να ακούμε μια πιο ε, μακροπρόθεσμη άποψη. Κάποιον δηλαδή που κοιτάζει πιο μακριά από τη στιγμή. Έχω να σχολιάσω πάνω σε κάποια προβλήματα που θίξατε. Πρώτα απ' όλα δημογραφική κρίση. Αναμφίβολα. Υπάρχει και έρχεται σε αντίθεση και θα συγκρουστεί με το κοινωνικό μας μοντέλο στο πολύ σύντομα. Όμως εγώ δεν πιστεύω ότι οι κυβερνήσεις είναι θύματα της έλλειψης ε, συνεκτικής αντίδρασης. Η εμπειρία μου είναι η εξής. Έχουμε πολλά προβλήματα για να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό ζήτημα σαν ένα κοινό ζήτημα. Γιατί πάντα μπαίνει η εθνική διάσταση και στο δημογραφικό. Και έτσι αντί να μιλάμε για το πρόβλημα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου ή το πρόβλημα της Ευρώπης, όχι μιλάμε για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν κάποιες ευρωπαϊκές πρωτεύουσε. Και ένα πρόβλημα που είναι διαρθρωτικό καταλήγει σαν ένα ε, ζήτημα εσωτερικής πολιτικής. Και οι ευρωβουλευτές μπαίνουν στην αμυντική θέση. Και αντί να χειρίζονται το ζήτημα όπως θα έπρεπε, μπαίνουμε στην ξύλινη γλώσσα και δεν βγαίνει τίποτα. Μα χρησιμοποιούν τελικά οι κυβερνήσει. οι οποίε εγώ πιστεύω ότι δεν είναι θύματα τη κατάσταση. αλλά, να το είπε πριν και ο συνάδελφος, οι κυβερνήσει μα οδηγούν σε, μια επαναθνικοποίηση των διαφόρων πολιτικών. Και όπως είπε και πριν ο συνάδελφος, πάντα λένε «Α, η Ευρώπη μας είπε να το κάνουμε αυτό». Μα δεν είναι αλήθεια. Και αυτό ισχύει με το δημογραφικό με τέτοια μοιοπία το κοινοβούλιο, το οποίο είναι διατεθειμένο φυσικά και να σώσει το οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο, δεν θα μπορεί. Γιατί, για άλλη μια φορά, βρίσκεται όμοιρος των εθνικών ιδεών των κυβερνήσεων και του Συμβουλίου. Το πρόβλημα της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης έχει και ένα ζήτημα νομιμοποίησης απέναντι στους πολίτες. Θα χρειαζόταν ένας χώρος όπου ζητήματα όπως είναι οι συντάξεις ή το κράτος ευημερία μακροπρόθεσμα να μην συνδέονται με την φορολογική ή πολιτική τα επόμενα δύο χρόνια. Γιατί αλλιώς συνδεκάτα, μη κυβερνητικέ οργανώσεις είναι κατά. Πώς λοιπόν να πετύχουμε τις ε, μεταρρυθμίσεις χρειάζεται και η καρδιά και το μυαλό των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτές ήταν κάποιες παρατηρήσεις που είχα να κάνω. Ο ε, Ευχαριστώ. Και σας κύριε Πρόεδρε και τον κύριο Γκονσάλες για την ενδιαφέρουσα ανάπτυξη του θέματος. Τρία σχόλια. Πρώτο, για το μέλλον. πριν από 20-30 χρόνια, πριν από την παγκοσμιοποίηση δηλαδή, μπορούσε κανείς να μαντέψει λίγο το μέλλον με κάποια σχετική βεβαιότητα. Αυτό τώρα είναι αδύνατον, γιατί είναι πάρα πολλές οι μεταβλητές. Και βεβαίως μια εκθετική αύξηση στον αριθμό των φόρεων που δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια σκηνή. Οικονομική, πολιτική, στρατιωτική, κοινωνική. Και αυτό καθιστά πολύ πιθανότερη την, το, πολύ πιθανότερο τον αλληλοσχετισμό μεταξύ των δυνάμεων αυτών να καταλήξει σε μια νέα κρίση όπως αυτή της Lehman Brothers. Και βεβαίως πολύ διαφορετικά από αυτά που έχουμε ζήσει ή τουλάχιστον εγώ από το 1945 και μετά. Υπάρχει λοιπόν μια διαρκής αλληλοσχέτιση. Η Κίνα. Εξετάζοντας την Κίνα απ' έξω, φαίνεται να είναι πολύ στέρεα. Στην πραγματικότητα, 25 έως 30% των μισθών της είναι κακή μισθή. Ε, ε, ε, συγγνώμη, τα, τα δάνεια. Είναι δάνεια τα οποία είναι επικίνδυνα. Μπορεί δηλαδή να καταρρεύσει κάποια στιγμή η κινέζικη οικονομία. Εν τέλει το ερώτημά μου είναι το εξή. Γιατί αυτό το ξυπνητήρι που χτύπησε για την Ευρώπη στην Κοπενχάγη δεν εισακούστηκε. Είμαστε πολύ λιγότερο σημαντικοί από ό,τι θεωρούσαμε. Δεν μας ακούει ο κόσμος. Γιατί αυτό δεν μας ξυπνά. Τώρα, δεύτερο, συμφωνώ με την ανάλυση σας σχετικά με το εθνικό κράτος, το κράτος έθνος, που για πολλούς είναι πολύ μεγαλύτερη πηγή ασφάλειας από ότι η Ευρώπη. Το αντίθετο από ότι πριν από 20-30 χρόνια. Η ερώτησή μου είναι πώς μπορεί κανείς να πείσει και τους εθνικούς πολιτικούς και τους πολίτες ότι ορισμένες τουλάχιστον κρίσεις επιλύονται πολύ καλύτερα και ασφαλέστερα στο ευρωπαϊκό επίπεδο από ότι στο επίπεδο του εθνικού κράτους. Και τρίτο σχόλιο είναι η ανώτερη εκπαίδευση. Εργάστηκα εγώ στην ανώτατη εκπαίδευση για πολύ καιρό. Η εμπειρία μου είναι ότι όταν σημειώνεται κρίση, οι περικοπές γίνονται κατά πρώτον λόγον εκεί. Δεν έχει ισχυρό πολιτικό σύστημα βάσης αυτή η ανώτατη εκπαίδευση. Τώρα, για αυτά που είπατε για την οικονομία που βασίζεται στη γνώση, και βλέπω πολλές χώρες να περικόπτουν τις δαπάνες στην ανώτατη εκπαίδευσή τους, νομίζω ότι κάθε χώρα μέλος έχει ενδιαφέρον να προωθεί την ανώτατη εκπαίδευση. Πώ θα το περάσουμε το μήνυμα αυτό. Ότι όλοι είμαστε ενδιαφερόμενα μέρη σε αυτή την υπόθεση και για την ενότητα εκπαίδευση όπω αυτή διεξάγεται στι άλλες χώρες. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την έκθεσή σας και για την παρουσίαση της έκθεσης αυτής που πάει ακόμα πιο μακριά. Ευτυχώς δεν είναι απλώς ενημέρωση. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω για το ρόλο της Μεσογείου, της Νότιας Μεσογείου κυρίως τα επόμενα δέκα χρόνια. Επηρεάστηκε από την κρίση, επίσης υπάρχει ο νέος ρόλος της Τουρκίας, μετά τα επεισόδια με τον ε, στόλο, με τα σκάφη δηλαδή. Η Κίνα έχει επίση νέο ρόλο. Νέες ενεργειακές συμφωνίες, καταπολέμηση της τρομοκρατίας, προετοιμασία για το κλίμα, περιβάλλον. Για την Μεσόγειο λοιπόν δεν νομίζω ότι έχουμε πει αρκετά και δεν κάνουμε αρκετά, ενώ από την άλλη μεριά της Μεσογείου μας περιμένουν, περιμένουν η, να φροντίσουμε και εμείς η Μεσόγειος να έχει να παίξει έναν ακόμα μεγαλύτερο ρόλο στο μέλλον. Ευχαριστούμε. Τελευταία παρέμβαση. Δύο, δύο ακόμα. Η κυρία Δικέιζερ πρώτη. Και, ο κύριο Μπρόγκ και μετά η κυρία Δικέιζερ. Πολύ σύντομα. Όχι, λέει ο πρόεδρο. Πρώτη Ποιος θέλει να μιλήσει πρώτος. Ο κύριος Μπρόνς θα μιλήσει πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον αυτά που είπε ο κύριος Γκονζάλης σχετικά με την ενιαία αγορά και τη δημιουργία του ευρώ και μία άλλη εξέλιξη, δεν τη σημειώσα αυτή, ότι όλα αυτά δημιουργήθηκαν από πάνω προς τα κάτω, είπε. Ενώ τώρα είναι αναγκαίο, λέτε, να κάνουμε την ίδια ένωση από κάτω προς τα πάνω. Ελπίζω να μην σας ε, παρανόησα. Είναι αυτό ακόμα ένα παράδειγμα της επιβλημένης ενότητας της Ένωσης. Απουσία ζήτησης, δηλαδή η ενότητα για να προχωρήσει θα πρέπει να προχωρήσει αντίστροφα, δηλαδή να υπάρχει ζήτηση για την, για την Ένωση και όχι το αντίστροφο. Ευχαριστώ. Ελπίζω να είμαι σύντομο. Πρόεδρο, σα ευχαριστούμε και η κυρία Δικέιζερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γκοντζάλα, πήγατε πολύ πιο πέρα από την έκθεσή σας σήμερα ευτυχώς προ όφελό μα. Θα ήθελα όμως στην τελευταία μου αυτή ερώτηση να μας πείτε κάτι για το πώς βλέπετε τη συνεργασία και την ανάπτυξη και το μέλλον τους στην Ένωση. Διότι στην έκθεση διαβάζουμε ότι πρέπει να υπάρχει μια πολιτική ανάπτυξη, σε εμπορική πολιτική έξυπνη εντό εισαγωγικών με δύσκολε αποφάσει φυσικά μετά τον κύκλο της Δόχα κλπ. Εφόσον όμως για όλα τα θέματα προχωρήσετε πέραν της έκθεση θα μπορούσατε και γι' αυτό να μας πείτε κάτι παραπάνω για το πώς εσείς βλέπετε το θέμα αυτό για την Ευρώπη, την ανάπτυξη και τη συνεργασία. Ευχαριστώ. <clears throat> Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος Γκονζάλες θα απαντήσει. Και πιστεύω ότι θα το κάνει σύμφωνα με την αρχική του εισαγωγή με ρεαλισμό και ελπίδα. Αυτός θα ήταν ο τίτλος που θα έβαζα εγώ στην ε, Δεν ξέρω όμως αν θα μπορέσω να πειθαρχήσω στο χρόνο που μας μένει. Ξεκινώντας από το τέλος, κύριε Μπρόντς. Αυτό που είπα, το είπα απόλυτα συνειδητά. Η Ευρώπη φτιάχτηκε ε, εξαιτίας της θέλησης κάποιων Ευρωπαίων ηγετών Έξι χώρες ήταν στην αρχή και επικεφαλής τους σκέφτηκαν ότι θα ήταν καλύτερο να τα βρούνε μεταξύ τους, να καθίσουν γύρω πάνω τραπέζι και αντί να ανταλλάσσουν ε, πυροβολισμούς, όπως έγινε δύο φορές τον 20ο αιώνα, να συμφωνήσουν. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες. Πάντως ήταν μια απόφαση, κατά τη γνώμη μου, των ευρωπαϊκών ελίτ της εποχής. Αυτή ουσιαστικά ανταποκρίθηκαν έτσι σε αυτό που ο κόσμος ήθελε, που ήταν ειρήνη. Όντως, η οικοδόμηση λοιπόν της Ευρώπης έγινε με πρωτοβουλία των επικεφαλής αυτών, κάτι όμως το οποίο δεν σημαίνει ότι δεν ανταποκρίθηκαν συγχρόνως και στην επιθυμία και τις επιθυμίες των περισσότερων των πολίτων, στην έκθεσή μας λέμε ένα σωρό πράγματα. Κάθε πράγμα που λέει κανείς μπορεί να τεθεί σε συζήτηση. Όλος παραδόξος όμως, όταν λέμε ότι η Ευρώπη θα έπρεπε να προσπαθήσει να μιλάει με μία φωνή στα διεθνή φόρα, όπως το Διεθνές Νομισματικό τομείο, η Παγκοσμία Τράπεζα κλπ. κλπ. Πάντα ακούμε ότι οι πολίτες δεν θα ανεχθούν να χάσουν κυριαρχία. Οπότε όλες οι αναλύσεις συμφωνούν με το ότι 80% των Ευρωπαίων πολιτών πιστεύουν ότι είναι πιο αποτελεσματικό να μιλάνε με μία φωνή στο, στην Κοπεχάγη, όπως κάνουμε και στην Τόχα, έτσι αλλά πρέπει να συμφωνήσουμε από πριν μεταξύ μας. Οπότε δεν φταίνε οι πολίτες. Οι πολίτες δεν διαφωνούν να παίρνουν οι επικεφαλείς τους μια πρωτοβουλία κτλ. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει το θέμα της κυριαρχίας. Και όταν εγώ λέω ότι πρέπει τώρα να φτιάξουμε τη συνέχεια από κάτω προς τα πάνω, το λέω γιατί εσείς εκπροσωπείτε τους Ευρωπαίους πολίτες πρώτα απ' όλα. Τώρα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα κύμα απαιτήσεων των πολιτών για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα είναι για να φτιάξουμε ακόμα περισσότερο μια Ευρώπη των πολιτών και δεν λέω ότι το υπόλοιπο οικοδόμημα έγινε σε αντίθεση με την πλειοψηφία των πολιτών. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Καφέ άλλο. Σας λέω ποια είναι η πεποίθησή μου. Οι χώρες που είναι λιγότερο υπέρ της Ευρώπης έχουν κοινωνικές πλειοψηφίες που γνωρίζουν ότι εκτός Ευρώπης κάνει πιο κρύο από ότι μέσα στην Ευρώπη. Και γι' αυτό και μένουν. Μπορεί να μην συμφωνούν με τη μία ή την άλλη πολιτική, αλλά να φύγουν δεν φεύγουν. Κανείς δεν θέλει να φύγει. Κανείς δεν θέλει να βγει. Γιατί αν πραγματικά θέλανε, πιστέψτε μου, θα είχαν φύγει. Ποιος θα τις εμπόδιζε. Εδώ δεν μπορούμε να εμποδίσουμε μια χώρα να μπλοκάρει, ας έχει 10 εκατομμύρια, την θέληση 15 για να επικυρωθεί μια συνθήκη. Η Ιρλανδία, εντάξει, ποτέ δεν ήθελε μέχρι τώρα να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα θέλει. Προφανώς. Ξαφνικά έχουν ενθουσιαστεί. Και υπάρχουν και άλλοι Ευρωπαίοι. Και αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι έγινε πιο ωραία, αλλά με το ότι τη χρειάζονται την Ευρώπη. Από αυτά που άκουσα και όλα μου δημιουργούν αίσθηση. Με τον ε, κύριο Γιάννη θα ξεκινήσω. Αν ξέρει ο κόσμος την έκθεσή μου. Όχι, δεν την ξέρουν. Αν αντέδρασε το Συμβούλιο που μου την ανέθεσε. Ναι. Υπάρχει ένα σημείωμα στα συμπεράσματα του Συμβουλίου που λέει ναι, λαμβάνουμε γνώση και ευχαριστούμε. Σε ποιο σιρτάρι τώρα θα μπει στη γραμματεία του Συμβουλίου. Αυτή η έκθεση δεν τολμάω να το σκεφτώ. Θα είναι στο πρώτο σερτάρι, στο τελευταίο, δεν ξέρω. Πολύ πιθανόν η προσπάθεια που δεν ήταν λίγη που κάναμε, να είναι μια προσπάθεια που θα οδηγήσει και αυτή στη μελαγχολία, μπορεί. Μα γι' αυτό προσπαθώ. Εγώ προσπαθώ να χτυπήσω το τύμπανο, να ακουστώ και εδώ ήρθα να σας εξηγήσω την έκθεση κάτω φασαρία, να ακουστώ. Μπα και μερικοί από εσά συμφωνήσουν μαζί μου, το δουν και αυτοί, ότι είμαστε σε μια πολύ περίπλοκη κατάσταση τώρα και ότι αν δεν αντιδράσουμε θα είμαστε με τους χαμένους. Τελεία και παύλα. Δεν το πιστεύουμε. Όταν το πιστέψουμε σε 20 χρόνια δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θα είναι πολύ αργά. Αυτή είναι η βαθιά μου πεποίθηση. Πολλοί με λένε απεσιόδοξο. Ε, τι θα κάνω. Εγώ σας λέω ότι είναι απεσιοδοξία με πολλή γνώση. Εγώ όμως δεν πιστεύω ότι είμαι ούτε απεσιόδοξος ούτε αισιόδοξο. Εξαρτάται τι θα κάνουμε με τη γνώση αυτή. Όταν λέτε ότι απ' έξω μας βλέπουν καλύτερα, ναι, πριν από ένα χρόνο, 50 μεγάλοι επιχειρηματίες μιλήσανε μαζί μου και τίποτα από όλα αυτά δεν λέγανε. Μου ζήτησαν 15 λεπτά να τους μιλήσω για το εξής. Ευρώπη, δύο τελείες. Μουσείο ή εργαστήριο. Κάντε το κι εσείς αυτό. Κάντε την προσπάθεια να απαντήσετε. Είμαστε μουσείο ή εργαστήριο. Και αν είμαστε μουσείο, τι μουσείο. Ήμασταν ένα πολύ καλό εργαστήριο ευημερίας, ε, ευημερίας προστασίας ε, των κεκτημένων Και ο Ομπάμα όταν θέλησε να κάνει μια μεταρρύθμιση, θέλησε να κάνει μια μεταρρύθμιση που έμοιαζε με αυτήν που είχαμε εμείς, την κατάσταση που είχαμε εμείς. Αλλά εμείς είμαστε σε μια κρίση. Φυσικά και οι Κινέζοι μας κοιτάνε με προσοχή για να μπορέσουν στο μέλλον να αποφύγουν τις κοινωνικές εντάσεις που δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε με ανακατανομή. Προφανώς και κοιτάνε και μας παρατηρούν να δουν, να μάθουν από μας. Αυτό που δεν κοιτάνε είναι την παραγωγικότητα των ώρα εργασίας. Για να το πούμε καθαρά. Εμείς πρέπει να το πούμε στους φίλους μας των συνδικάτων. Αυτό δεν προσπαθούν να το αντιγράψουν από μας. Όχι. Αυτό λοιπόν που με απασχολεί είναι ότι αν πάνω σε αυτό δεν έχουμε να πούμε τίποτα, δεν έχουμε να πούμε τίποτα και για τη διατήρηση του κοινωνικού μας μοντέλου. Πρέπει να είμαστε λοιπόν συνεπείς με τους αυτούς μας. Εγώ δεν θέλω καμιά θέση, έτσι. Να ξέρετε. Κάθε άλλο. Θέλω να ελευθερωθώ από αυτό. Αλλά δεν μπορώ να κρύψω αυτά που έχω να σας πω. Ότι μας βλέπουν καλύτερα απ' έξω. Ναι, Λατινική Αμερική και άλλες χώρες, οι οποίες ονειρεύονται ένα μοντέλο σαν το δικό μας. Φυσικά. Και εγώ είμαι ερωτευμένος με αυτό το κοινωνικό μοντέλο, αλλά το θέλω για τον 21ο αιώνα, όχι για τον 20ο. Αν δεν το δούμε αυτό, οι κυβερνήσεις θα προχωράνε μέσα στην κρίση, θα αντικαθίστανται από τις επόμενες κυβερνήσεις και ούτω καθεξής θα αλλάζουν οι κυβερνήσεις, η προηγούμενη θα ξανάρχεται και ούτω καθεξής. Σας είπα και εγώ για τη διακυβέρνηση, το άκουσα και από πολλούς από εσά. Οι προχωρημένες δημοκρατίες αντιμετωπίζουν αυξανόμενα προβλήματα διακυβέρνησης. Και γι' αυτό και πριν σας έδωσα για παράδειγμα την Καλιφόρνια. Δεν ήθελα να μιλήσω γενικά για τον Ομπάμα, το περιθώριο ελιγμών του περιορίστηκε πολύ. Η εντολή του ήταν ε, τύπου Ρούσβελ. Και όχι Κάρτερ. Εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα τον Κάρτερ ως προσωπικότητα, όμως όχι το αποτέλεσμα. Υπάρχει ένα πρόβλημα διακυβέρνησης, σοβαρό, στις προχωρημένες δημοκρατίες, στις προηγμένες δημοκρατίες. Και αυτό έχει να κάνει με τους νέους παράγοντες στις μεγάλες χώρες. Η ΑΣΕΑΝ, η ομάδα ΑΣΕΑΝ που συνεδριάζει αυτές τις μέρες στις Βρυξέλλες, σε ποιον θέλει να μοιάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στα θετικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι στα στραβά, και έχει μία μόνιμη ομάδα εργασίας εδώ και καιρό που παρατηρεί τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να δούνε τι θα κρατήσουν και τι θα πετάξουν. Υπάρχουν λοιπόν νέοι ε, φορείς σε διεθνές ε, επίπεδο από νέες χώρες που δεν πρέπει να παραβλέψουμε και που μερικές φορές δεν θέλουμε να λάβουμε υπόψη μας. Τόσο το χειρότερο για μας. Με τον πρόεδρο του Ιράν δεν θα υπάρξει συμφωνία με την Τουρκία, η Τουρκία μάλλον ή η Βραζιλία θα υπογράψουν συμφωνία. Εκνευρισμό δημιουργεί κάτι τέτοιο. Όμως έξι μήνες χωρίς αυτές τις χώρες. Αν αποφασίσει να υπογράψει την ίδια συμφωνία, την ίδια, με τους ίδιους όρους. τι θα έχει γίνει με τη Βραζιλία και την Τουρκία, θα μας έχουν προλάβει. Θα έχουν υπογράψει τη συμφωνία που το Ιράν μπορεί να έχει πει ναι στην Βραζιλία και την Τουρκία και να πει μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανησυχία μου είναι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα διακυβέρνησης στις προηγμένες δημοκρατίες εξαιτίας της εμφάνισης πολλών παραγόντων που δεν είναι οι παραδοσιακοί, ούτε τα παραδοσιακά πολιτικά κόμματα. Νέοι παράγοντες λοιπόν που δεν ξέρουμε πώς να τους λάβουμε υπόψη μας για να συνεισφέρουν υπέρ μιας καλής διακυβέρνησης. Αυτή η καταπληκτική ιδέα που είναι η πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών που θα οδηγήσει σε νέους νόμους οφείλεται στην κρίση διακυβέρνησης, όχι Ευρωπαίου, συγγνώμη, η αντίστοιχη στην Αμερική, στην Καλιφόρνια, οδήγησε στην κρίση στην Καλιφόρνια. Αν δεν θέλουμε να το δούμε αυτό, θα βρεθούμε μπροστά στο πρόβλημα αργότερα. Είπαμε λοιπόν για τα δημογραφικά. Δεν φτάνει να πω ότι όλοι είμαστε σε ένα παιχνίδι μεταξύ της εθνικής διάστασης και της ευρωπαϊκής διάστασης. Ζητάμε από την Ευρώπη να δώσει απαντήσεις σε προβλήματα εθνικού επίπεδου. Λειτουργία οικονομικού συστήματος και έλεγχος. Να, αυτό δεν μπορεί να το λύσει από μόνη της καμία χώρα. Ούτε καν ολόκληρη η Ευρώπη δεν μπορεί να το λύσει. Μόνο σε συμφωνία με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Μόνο ε, στη κυκλοφορία κεφαλαίων, όχι μόνο δικών μας και άλλων, μόνο εκεί μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάποια ηγεμονία. Αλλά ακόμα και έτσι το 80% της αγοράς κεφαλαίων περνάνε από τρεις χώρους. Όχι όμως η ρύθμιση. Η ρύθμιση πρέπει να είναι μια πρόταση τακτοποιημένη, μακάρι να είναι Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης. Που να δεχτούν οι διάφοροι δημοσιονομικοί οργανισμοί. Έχουμε λοιπόν πολύ σοβαρά προβλήματα διακυβέρνησης και δεν τα σκεφτόμαστε αρκετά. Νομίζουμε Λέμε ότι η δημοκρατία πρέπει να είναι πιο ανοιχτή, η τεχνολογία να επιτρέπει πρόσβαση σε όλα, αλλά όχι στις αποφάσεις. Και έτσι καταλήγουμε στα προβλήματα διακυβέρνησης. Στη Wall Street, ο Ομπάνα όταν μίλησε για τη δημοσιονομική ε, μεταρρύθμιση, ήταν τέλεια η ομιλία του εκεί τέλεια. Και αυτό που ζήτησε τελικά από τη Wall Street για να τον βοηθήσουν υπέρ της μεταρρύθμισης ήταν αντίφαση. Ε, βοηθήστε να μεταρρυθμίσουμε τους μηχανισμούς από τους οποίους εσείς έχετε μάθει να κερδίσετε πολύ χρήμα. Δεν τους το είπε έτσι. Βοηθήστε με να αποφύγω τις αντιστάσεις του Κογκρέσου. Εσείς μπορείτε να με βοηθήσετε σε αυτό, τους είπε. Ε, δεν θα το βοηθήσουν. Σιγά μην το βοηθήσουν. Δεν είναι δυνατόν. Λέω λοιπόν πάλι. Χάνουμε, πάμε πίσω, χάνουμε τη σύνδεση με την πραγματικότητα. Υπήρχε ένας τίτλος «Το μέλλον δεν είναι αυτό που ήτανε». Βιβλίο από τον προηγούμενο αιώνα. Πολύ καλό ένας νέος παράγοντας που έχει μπει στη ζωή μας και στη γενιά μας είναι η εκθετική αύξηση της έλλειψης προβλεψιμότητας. Παρόλο που έχουμε τεράστια επικοινωνία μεταξύ μας. Ο άνθρωπος είναι ιστορικό «ον». Μαθαίνει από το παρελθόν, είτε στο πανεπιστήμιο, είτε στην πόλη, στο χωριό μαθαίνει από το παρελθόν. Τώρα τα παιδιά διδάσκουν στους μεγαλύτερους πώς να χειρίζονται αυτά τα διαβολικά μηχανήματα που θα έλεγε η Εκκλησία το 19ο αιώνα, που είναι ηλεκτρονικοί υπολογιστέ Σε μια γλώσσα ψηφιακή. Ο άνθρωπος που είναι ιστορικό «ον» αποδομείται. Νιώθει κάποια αγωνία. Δεν νιώθει άνετα. Γιατί καταλαβαίνει ότι αυτό που ήξερε δεν θα είναι. Και ο κώδικας που χρησιμοποιούσαμε μέχρι τη δικιά μας γενιά για να ερμηνεύσουμε τα γεγονότα δεν μας χρησιμεύει πια. Αλλάζει ο κόσμος. Μάλλον δεν αλλάζει. Άλλαξε ο κόσμος. Και εμείς καθόμαστε και τσακωνόμαστε για ένα μέλλον. Για, ένα, για να κερδίσουμε ένα μέλλον το οποίο έχουμε ήδη πίσω μας. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται κατάλληλη διακυβέρνηση η Ευρώπη και είναι τόσο σημαντικό αυτό. Το λέω αυτό και στις κυβερνήσεις και στις αντιπολίψεις. Λένε η Ευρώπη μας υποχρεώνει. Μα ποια είναι αυτή η Ευρώπη. Εγώ δεν την ξέρω την κυρία Ευρώπη. Και όταν βλέπω τις διαδηλώσεις κατά της κρίσης, ε, πρέπει να ξέρουμε πού πάμε και διαμαρτυρόμαστε. Η Ευρώπη είναι το άλοθη τελικά και των κυβερνήσεων και της αντιπολίτευσης σε κάθε χώρα. Υπάρχει κάτι που πληρώνει τώρα πια ο κόσμος και το οποίο δεν το επιβάλλει κανένας από όλους αυτούς. Το επιβάλλουν οι αγορές. Η αντιπολίτευση λέει «Α, όχι, δεν θα το είχατε κάνει αν δεν σας υποχρέωναν οι Βρυξέλλες». Μα τελικά δεν βλέπει ο κόσμος πέρα από τη μύτη του. Αν 27 αποφασίζουν να κάνουν κάτι με το οποίο δεν συμφωνούν, που είναι μία ε, πολιτική εξυγένση των δημοσιονομικών, ε, τελείωσε. Ποιος επιβάλλει σε ποιον. Όταν αποφασίζουν για ένα ε, μια συμφωνία σταθερότητας και όταν υπογράφουν στο Συμβούλιο υπογράφουν και αυτό σημαίνει ότι και 27 συμφωνούν. Δεν μπορεί λοιπόν να έρχεται ο ένας ή ο άλλος και μετά να λέει «Α, μας το έχουν επιβάλει οι Βρυξέλλες». Έπειτα, περικοπές. Εύκολο να τις κάνει κανείς την εκπαίδευση. Και όμως, είναι λυπηρό που είναι έτσι. Είπατε έπειτα για την Μεσόγειο και συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου ανάπτυξη κλπ. Λοιπόν, Νότιο Μεσόγειο. Το 1995 πολύ χάρηκα που ξεκίνησε στην Βαρκελόνη μια πολιτική ειδικά για την Νότια Μεσόγειο. Πέρασε τόσο καιρό όμως που... Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχει γίνει τίποτα. Είχαμε αποφασίσει ήδη από πριν στη Γαλλία για τη χρηματοδότηση της πολιτικής αυτής. Και είχα πει στον Κολ τότε, για να τον καθησυχάσω, ότι ο προπολογισμό θα ήταν το 70% του προπολογισμού που πήγαινε στις διαθροτικές πολιτικές που προέβλεπαν τη διεύρυνση προς τις χώρες της Ανατολικής τότε Ευρώπης. Δεχτήκαμε αυτή την πολιτική με την Προεδρία του τότε Γάλλου Προέδρου. Υπήρχε λοιπόν το δημοσιονομικό πακέτο. Υπήρχαν τα λεφτά. Και μετά η συμφωνία. Η συμφωνία δεν λειτουργήσε, όχι. Γιατί, Γιατί κανένα δεν τη έδωσε συνέχεια. Κανεί. Τώρα έχουμε μια νέα έκκληση. Μια νέα πολιτική για τη Μεσόγειο. Αλλά και πάλι. Κανένας δεν δίνει συνέχεια. Τι γίνεται λοιπόν με τη Μεσόγειο η θεωρία των μεγάλων συνόλων που δεν πρέπει να υποτιμάει κανείς. Στην Κίνα όταν πήγα πριν από 25 χρόνια, ο Τζοπίν μου είπε Πώς είσαστε στην Ευρώπη. Ήμασταν πριν τη διεύρυνση. Του είπα πόσα εκατομμύρια ήμασταν. Και μου λέει, καλά, τόσο λίγοι είσαστε, δεν μπορείτε να συμφωνήσατε». Αλήθεια σα, λέω, έτσι μου είπε. Με το συλλογή είσαστε. Ε, συμφωνήστε τέλο πάντων μεταξύ σα. Λοιπόν, στη θεωρία αυτή των συνόλων που φτιάχνονται στον κόσμο, Ηνωμένε Πολιτείε Καναδά, Μεξικό, κοινωνία, έτσι η Κίνα μάλλον από μόνη της φτάνει, δεν χρειάζεται κανένα για να φτιάξει σύνολο, παρόλα αυτά έχει την ΑΣΕΑΝ και θέλει να πρωταγωνιστεί βέβαια. Λοιπόν, σε αυτή τη θεωρία των συνόλων, με 50 εκατομμύρια και αν βάλουμε και την Τουρκία και αν βάλουμε και την Μεσόγειο, για σκεφτείτε, το σύνολο αυτό είναι λιγότερο από την Κίνα. Και έχουμε αυτά που λείπουν από τον Νότο και αυτά που λείπουν από το Βορρά. Πρέπει να είμαστε λιγάκι εγωιστικά ευφυείς. Και δεν μιλάω εδώ πέρα για αλληλεγγύη. Έχουμε καταχραστεί αυτή τη έννοια. Δεν θα ήταν λογικό να τα βρούμε μεταξύ μας. Να αναλύσουμε πού είμαστε συμπληρωματικοί μεταξύ μας. Ξέροντας ότι δεν μπορούμε να κρατήσουμε τον κατώτατο μισθό περνάντας από την άλλη μεριά του Γιβραλτάρ. Δεν είναι δυνατόν ο ελάχιστος μισθός μας να μπορεί να είναι πάνω από το μέσο όρο του μισθού εκείνων που είναι από την άλλη μεριά του Γιβραλτάρ και όταν τον έχουν αυτό το μισθό. Δεν πέρασαν μια κρίση σαν και εμάς, οπότε γι' αυτό είπα και στην αρχή όταν ξεκίνησα και το έχω πει πολλές φορές μέχρι τώρα. Δεν θα ήταν καλό να καθίσουμε να σκεφτούμε λίγο για την Ευρώπη με το εξή ερώτημα. Γιατί μας μας πλήττει η κρίση οικονομική περισσότερο από ό,τι τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ασία, τη Λατινική Αμερική κτλ. Γιατί η απάντηση είναι σχετικά εύκολο να τη διατυπώσει κανείς, αλλά πώς να διορθώσει την κατάσταση. Γιατί η κρίση βρήκε μια Ευρώπη που βρίσκεται 10-12 χρόνια πίσω σε σχέση με τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις που θα έπρεπε να έχει εφαρμόσει. Και γι' αυτό είμαστε ευάλωτοι. Και γι' αυτό μας έπληξε πιο πολύ εμάς η κρίση, γιατί είμαστε πιο τρωτοί. Ένα από τα καλύτερα πράγματα που έχουμε στην συνεργασία για την ανάπτυξη. Είναι και αυτό το λέω πάντα για να μην έτσι σαν αστείο, για να ελαφρύνω λίγο την ατμόσφαιρα. Μερικές φορές η Ευρώπη πιστεύει ότι αν δεν έχουμε sex appeal, δεν μπορούμε να διορθώσουμε τα πράγματα. Όχι, δεν είναι έτσι. Το εμείς χρειαζόμαστε ένα check για να μπορέσουμε να κερδίσουμε έδαφος. Και η Ευρώπη πρέπει να έχει βάρος, γιατί εμείς πιστεύουμε στις αξίες μας και η συνεργασία με τον έξω κόσμο είναι ένα στοιχείο. Κάτι πρέπει να αλλάξουμε. Κάποιες χώρες έχουν ήδη ξεκινήσει. Πρέπει να αλλάξουμε τη συνεργασία για να ξέρουμε οι χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε πώς μπορούν να τροποποιήσουν τα δικά τους οικονομικά συστήματα για να ενταχθούν στην κοινωνία του 21ου αιώνα της οικονομίας της γνώσης. Πολλές χώρες της Βόρειας Ευρώπης το κάνουν. Και το διαπιστώνω αυτό. με χρήματα που πηγαίνουν στην καινοτομία. Κάτι το οποίο θα βοηθήσει πολύ στο μέλλον και επενδύουν και σε χώρες με τις οποίες εμείς συνεργαζόμαστε από την Αφρική και αλλού. Η συνεργασία μας είναι από τις υψηλότερες όλο τον κόσμο, συγκριτικά. Η Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία κάποτε καθόριζαν την τιμή των πρώτων υλών, γιατί είχαν ολιγοπόλιο ζήτησης. Εμείς καταναλώνουμε, οπότε τόσο θέλουμε εμείς τον καφέ, τόσο θέλουμε το χαλκό και το καθεξής. Και αφού εγώ είμαι η βιομηχανία που τη χρειαζόσαστε εσείς και η βιομηχανία θα κοστίζει όσο λέω εγώ. Οπότε εμείς καθορίζαμε την τιμή των πρώτων υλών και την τιμή της μεταποίησης. Ε, αυτή η ιστορία τελείωσε, έληξε. Στην Τόχα λοιπόν μπορεί να γίνει ό,τι θέλετε. Αλλά οι σχέσεις που συζητιώνται στην Τόχα των συναλλαγών δεν περνάνε από την αγορά ε, της, των πρώτων υλών με τιμές που εμείς αποφασίσαμε, ούτε από τη ΣΥΤΗ. Η ζήτηση δεν είναι πια η ζήτηση των αναπτυγμένων δυτικών χωρών που καθορίζουν την τιμή των πρώτων υλών και της μεταποίησης. Όχι. Τώρα η Κίνα είναι και η βιομηχανία και η μεταποίηση και μερικές φορές και η Λατινική Αμερική. Οι επενδύσεις εκεί πάνε λοιπόν. Επιπλέον αγοράζουν και δικές μας βιομηχανίες. τις καλύτερες, τις πιο καλές. Τώρα έχουμε την κρίση του σίδηρου. Τι θα πούμε, στον Ταβινιό να κάνει την ε, μεταρρύθμιση. Για να δούμε τι θα γίνει με το σίδηρο της Ευρώπης. Όλα αυτά πρέπει να καθίσουμε να τα σκεφτούμε, γιατί η Ντόχα σε σχέση με τη συνεργασία έχει πολύ διαφορετική σημασία. Λέμε για πράγματα που έγιναν στις διαπραγματεύσεις ε, στις Ντόχα και οι άλλοι από τη Βραζιλία και τα λοιπά συνεχίζουν να συζητάνε στην Ντόχα για τα πράγματα για τα οποία έχουν ε, δίκιο. Εμεί για τα πράγματα που δεν έχουμε δίκιο θέλουμε επίση να συνεχίσουμε να συζητάμε στην Τόχα για συμφέροντα τα οποία ήταν του παρελθόντο και δεν είναι ούτε του παρόντο ούτε του μέλλοντο. Άσε τι γίνεται όταν πλησιάσει κανεί τι εθνικέ πραγματικότητε. Γιατί κυριαρχούν οι εθνικές διαστάσεις, η εθνική διάσταση. Γιατί. Γιατί εκεί κερδίζει και χάνει η εξουσία και κερδίζει και χάνει η εξουσία μερικές φορές μιλώντας κατά της μετανάστευσης ή κατά το διαπραγματεύσεων στην Τόχα. Έτσι κερδίζει ψήφους. Που θα καθορίσουν αν θα έχει ή δεν θα έχει πλειοψηφία μετά τις εκλογές. Δεν λύνει όμως το πρόβλημα. Κερδίζει τις εκλογές. Αντί τις κέρδισε. Και το πρόβλημα δεν το έχει λύσει. Και γι' αυτό εγώ θα ήθελα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βλέπει τα πράγματα ευρύτερα να συμφωνήσει σε ένα πρόγραμμα τεσσάρων προτεραιοτήτων που να δουλέψει όμως. Μακάρι. Τότε εγώ ευχαρίστω να έρθω όσες φορές θέλετε να σας τα πω, να σας τα ξαναπώ και να βοηθήσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πρόεδρε Γκοζάλες, για το χρόνο που μας δώσατε. Και μου άρεσε πάρα πολύ τα τελευταία λόγια που κλείσετε και που γράψετε και στην έκθεσή σας. Αλλά θέσετε μερικά μικροπροβλήματα, θεωρητικά ίσως. Ούτε κι εγώ έχω συναντήσει την Ευρώπη στο δρόμο μου. Αλλά ούτε και τα κράτη τα έχω συναντήσει στο δρόμο. Ωστόσο, οι πολίτες έχουν ζήσει διάφορες καταστάσεις με τα γκούλακ, με το Χίτλερ κλπ. Ίσως νιώθουμε την Ευρώπη στο πνεύμα της ε, αδελφότητας που μας ενώσει, ενώνει, στην ελπίδα που μας ενώνει. Πιστεύω λοιπόν ότι οι τελευταίες λέξεις του γραπτού σας κειμένου δίνουν απάντηση στο ερώτημα που επαναλαμβάνω θέσατε Ευρώπη. Ε, μουσείο ή εργαστήριο. μουσείο θα έλεγα και μνήμη. Στο εργαστήριο είναι ένα σχέδιο, ίσως και υπάρχει μία λέξη. Αποστολή και τη γράψετε στο κείμενό σας. Αυτή η αποστολή απαιτεί πολιτικό θάρρος και συλλογική φιλοδοξία, πραγματισμό, ρεαλισμό και αίσθηση των ιδεωδών και να δοθεί μάχη εσωτερικά και εξωτερικά. Σας ευχαριστούμε. Gracias, presidente. Me voy a vivir a Florencia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 Allora possiamo continuare. Passerei al... Να συνεχίσουμε λοιπόν. Σημείο 6 της της διάταξης. Αποκινούμε το 7. Το αφορά την αναφέρεση της συμφωνίας πλαίσιο για τη σχέση Ευρωκοινοβούλιο και Κομισιόν. Εισηγητής Ράντζελ. Υπάρχουν τροπολογίες, DAF, του εισηγητή. Και τέσσερις τροπολογίες των συναδέλφων Ντάφ και Young. Παρακαλώ τον συνάδελφο Ράντζελ να μας εξηγήσει τι συνιστά για τις ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτη παρατήρηση. Αυτή η συμφωνία πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό επίτευγμα για το Κοινοβούλιο. Μερικές λεπτομέρειες της έκθεσης και των τροπολογιών να μην είναι τόσο σημαντικές. Να το συγκρίνουμε με το, στη σημασία αυτής της συμφωνίας πλαίσιο πρώτη μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Στηρίζεται στη συνθήκη σε συγκεκριμένο άρθρο. Τώρα εδώ έχουμε δύο ειδών τροπολογίες. Τροπολογία στην έκθεση που αλλάζει τους κανόνες διαδικασίας με τις συνέπειες της συμφωνίας πλαισίου στις δικές μας εσωτερικές διαδικασίες και κανονισμό εκεί δεν θα έχουμε προβλήματα τεχνικές είναι λεπτομέρειες μόνο για να έχουμε μια νομικά πιο σαφές τοπίο και μορφή έκφρασης των διαφορετικών συνεπειών της Συμφωνίας Πλαίσιο. Μερικές τροπολογίες που προτείνει ο Στάφος Νταφ από κοινού καταλήξαμε σε συμβασμό στα σημεία 17, 18, τροπολογίσμα 17, 18 και 19 διότι ο στόχος μας ήταν ο ίδιος. Απλώς η διατύπωση ήταν διαφορετική. Προσπαθήσαμε λοιπόν να πετύχουμε ένα συμβασμό. Έχουμε λοιπόν τρεις συμβαστικές τροπολογίες όσον αφορά τον κανονισμό σε σχέση με τις αρχικές προτάσεις 17, 18 και 19. Οι τροπολογίες ε, στην έκθεση. Συμφωνώ με την τροπολογία 4. Άντρου Νταφ. Την τροπολογία 3 του συναδέλφου Ντε Γιόγκ. Προτιμώ το κείμενο, είναι πιο σαφές, το αρχικό κείμενο. Και έχουμε και την τροπολογία 1 και 2 θα πρέπει να τις σκεφτούμε λίγο παραπάνω. Τροπολογίες του Σανδέφ Αντριντάφ. Η μία είναι πιο εύκολη. Οι δύο. Εκεί που ο συνάδελφος προτείνει όταν αναφερόμαστε ώστε να υπάρχει τακτικός διάλογος μεταξύ του Πρόεδρου της Κομισιόν και του Πρόεδρου του Κοινοβουλίου να πούμε χωρίς αυτό να μειώνει το ρόλο των προέδρων των σε, στα πλαίσια της δημοσιονομικής διαδικασίας. Νομίζω ότι αυτό δεν προσθέτει τίποτα. Ούτε καλό ούτε κακό είναι. Πάντως δεν προσθέτει τίποτα κάτι γνώμη μου. Γιατί αν δούμε τη συμφωνία πλαίσιο, το κείμενο, είναι σαφές ότι η διάσκεψη των Προέδρων κρατάει τις εξουσίες της. Άθικτες. Για να μην πω ότι έχει περισσότερες εξουσίες από ό,τι πριν. Ειλικρινά λοιπόν πιστεύω ότι δεν είναι αναγκαία αυτή η τροπολογία. Φυσικά δεν θέλουμε να μειώσουμε το ρόλο της διάσκεψης των Προέδρων. Ούτε στο γράμμα της συμφωνίας, ούτε στο πνεύμα της συμφωνίας ταιριάζει αυτό. Εγώ προτείνω αποχή. Αυτό που θα έπρεπε να σκεφτούμε όμως Να είμαστε προσεκτικοί με άλλα λόγια. Είναι η τροπολογία 1. Είναι αιτιολογική σκέψη. Λέμε, λαμβάνοντα υπόψη τη συνθήκη τη Λαμβάνωση θέτω Κοινοβούλη, ό,τι ισότιμη θέση με το Συμβούλιο στη συνήθεια νομοθετική διαδικασία και σε θέματα προπολογισμού και ενισχύει το ρόλο του στην εξωτερική πολιτική της Ένωσης με εξαίρεση το ρόλο του σε θέματα κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Ο Στέφος Νταφ προτείνει να διαγράψουμε την τελευταία φράση με εξαίρεση. Είναι αναγκαία αυτή η φράση. Γιατί λέμε ισότιμη θέση με το Συμβούλιο. Δεν πρέπει να έχουμε ισότιμη θέση σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Αυτό είναι σαφές με βάση τις συνθήκες και με τη Συμφωνία Πλαίσιο. Δεν πρέπει να φύγει αυτή η φράση. Να διαβάσουμε την έκθεση. Θα δούμε ότι υπάρχει πολύ ισχυρή θέση του Κοινοβουλίου όσον αφορά την εξωτερική διάσταση. Το Κοινοβούλιο έχει ισχυρή θέση. Οπότε, τι χρειάζεται να το ενισχύσουμε αυτό στην αιτιολογική σκέψη. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για ισότιμη θέση ως προς το Συμβούλιο σε θέματα νομοθετικά και προϋπολογισμό. Πρότασή μου λοιπόν είναι να καταψηφίσουμε την τροπολογία 1. Αυτή είναι η προσωπική μου θέση. Αδιαμφισβήτητα η έκθεση ορίζει και υποστηρίζει τη θέση του Κοινοβουλίου στον έλεγχο των εξωτερικών σχέσεων της εξωτερικής διάστασης της ευρωπαϊκής πολιτικής. Ακόμα και με μια πρώτη ματιά το αντιλαμβάνεται κανείς αυτό. Και αυτό είναι άμεσο αποτέλεσμα της διαπραγματευτικής ομάδας στη συμφωνία πλαίσιο. Δεν είναι μόνο θέση του εισηγητή. Είναι απορρέει από την εντολή που δόθηκε στη διαπραγματευτική ομάδα. Δεν κερδίζουμε τίποτα διαγράφοντας αυτή τη διευκρίνηση. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να καταψηφιστεί η υπαριθμόν 1. Πάντως, επαναλαμβάνω, το σημαντικό είναι ότι έχουμε την έκθεση τη συμφωνία πλαίσιο, γιατί η συμφωνία πλαίσιο είναι σημαντική, όχι η έκθεση. Κύριε, μεγάλο επίτευγμα για το Κοινοβούλιο που προσπαθεί συνεχώς να ενισχύσει τη συνταγματική του θέση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Θέλει κανείς να μιλήσει, ιδιαίτερα από αυτούς που πρότειναν τροπολογίες. Ο κύριος Ντάφ έχει το λόγο. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Πάουλο Ραντζέλ για την εισαγωγή που έκανε στο θέμα και στις τροπολογίες μου με τόσο ενδελεχή τρόπο. Ωστόσο, η Επιτροπή Συνταγματικών θα πρέπει να τοποθετηθεί κριτικά επί των επί της εκβάσεως των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επί των κανόνων διαδικασίες δέχομαι αυτά που λέει για το 17 και το 19. Συμφωνώ. Για την έκθεση η τροπολογία 2 Ας μην είμαστε αφελείς. Η συμφωνία πλαίσιο προτείνει τελείως διαφορετική πρακτική από την ισχύουσα, προτείνοντας ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου να συμμετέχει σε συνεδριάσεις του Σώματος των Επιτρόπων. Αυτό ενδέχεται να είναι ακίνδυνο, αλλά και ενδέχεται να αποτελέσει ωστόσο παραβίαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών και θα μπορούσε να επιτρέψει σε κάποιον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, ο οποίος δεν θα είχε κανένα δισταγμό, να παρεμβαίνει σε διαδικασίες προϋπολογισμού ή θεσμικές που προβλέπονται από τη συνθήκη κινούμενος παράλληλα εκτός της εντολής που του έχει δοθεί από την διάσκεψη πρόεδρων πολιτικών ομάδων. Βρίσκω λοιπόν ότι είναι σημαντικό ευγενός μεν να θυμίζουμε ωστόσο ότι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου περιορίζεται στα όσα μπορεί να πράξει εάν εν τέλει συμμετέχει σε συνεδριάσεις της Επιτροπής. Χωρίς να θέλω να βάλω κατά της ακαιρεότητας του παρόντος πρόεδρου Μπούσεκ, του οποίου συμπεριφορά είναι άψογη, αλλά δεν μπορεί να είναι πάντοτε και απόλυτα εξασφαλισμένο ότι ο διάδοχός του ή η διάδοχή του θα είναι και αυτή άψογη. Για την πρώτη τροπολογία νομίζω ότι πρέπει όπως πάντοτε να σεβαστούμε την λογική της συνθήκη της Λισαβόνας η οποία συγχωνεύει την ΚΕΠΑ και τις άλλες εξωτερικές δράσεις της Ένωσης. Γι' αυτό λόγο γίνεται άλλωστε και αυτό επιτύχαμε με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και θα ήταν λάθος να τις ξεχωρίσουμε. Νομίζω επίσης ότι μάλλον δεν αληθεύει το ότι δεν έχει αυξηθεί, δεν έχει ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου από την συνθήκη στην ΚΕΠΑ. Και τέλος, εάν ήταν αληθές αυτό, θα ήταν παράλογο να βγει το ίδιο το Κοινοβουλίο να το πει. Ο Παύλο Ραγγέλ λέει ότι μιλεί για ισότιμη βάση Κοινοβουλίου και Συμβουλίου στο προκείμενο θέμα. Ε, εγώ δεν το βλέπω έτσι στο σχέδιο δηλαδή της αιτιολογικής σκέψης. Μιλεί για ισότιμη βάση για θέματα νομοθετικά και δημοσιονομικά, σωστό αυτό, αλλά συνεχίζει λέγοντας ενισχύει τον ρόλο του σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Και αυτό σωστό είναι. Δεν λέει ότι το Κοινοβούλιο είναι σε ισότιμη θέση στην εξωτερική πολιτική ή στην ΚΕΠΑ. Για τους λόγους που ανέφερα λοιπόν, βρίσκω ότι είναι σημαντικό να παραμείνουμε μέσα στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε την προσπάθεια συνεργασίας μεταξύ Ευρωβουλής και Εθνικών Κοινοβουλίων στον χώρο της και πά κάτι το οποίο νομίζω ότι θα μας αναγκάσει κιόλας να λάβουμε υπόψη και να ενισχύσουμε το ρόλο του Κοινοβουλίου. Εσείς κύριε Ρομέρο που είστε επικεφαλής του, ε, της νομικής υπηρεσίας της Κομισιόν. Από Πλευρά Κομισιόν συμφωνούμε με τα όσα διαβεβαίωσε ο κύριος Ραονζέλ που μίλησε για επίτευγμα όταν μίλησε για την συνθήκη, για τη συμφωνία μάλλον πλαίσιο. Είναι πραγματικά εξαιρετικό το αποτέλεσμα και υπέρ των δύο θεσμικών οργάνων. Εμεί είμαστε ικανοποιημένοι από τις συστάσεις που λαμβάνει στην έκθεσή του ο κύριος Ραντζέλ, δηλαδή να εγκριθεί η συμφωνία πλαίσιο. Από πλευρά Κομισιόν θα τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας και θα εφαρμόσουμε την συμφωνία όπως την ε, συμφωνήσαμε μαζί σας. Ωστόσο, επισημαίνω, κύριε Πρόεδρε, το γεγονός ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής στην πράξη της Συμφωνίας Πλαισίου θα γνωρίζετε ότι για ορισμένους η συμφωνία πλαίσιο είναι ήδη υπερβολική. Όθεν υπάρχει κίνδυνος προσφυγής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ακόμη περισσότερο κίνδυνος προσφυγής κατά των πράξεων που θα ε, εγκριθούν κατ' εφαρμογή της συνθήκης πλαισίου. Άρα να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της και σε ό,τι αφορά την τήρηση απολύτως των πλαισίων των αρμοδιοτήτων που επιβάλλει η συνθήκη ε, πλαίσιο. Η Κομισιόν δεν θα μπορέσει να συμφωνήσει με ορισμένε εκ των ερμηνών που περιλαμβάνονται στην έκθεση Ραντζέλ που για μας υπερβαίνουν τα όρια του συμφωνημένου κειμένου της Συμφωνίας Πλαισίου. Για να αποφευθεί η αδίποτε ασάφεια και να είμαστε προετοιμασμένοι απέναντι σε οποιαδήποτε ενδεχόμενη προσφυγή, θα πρέπει οι ερμηνείες αυτές να θεωρηθούν ως πολιτική, μακροπρόθεσμα πολιτική στόχη του Κοινοβουλίου, αλλά είναι θεμελιώδους σημασίας και μιλώ καθαρά νομικά, είναι σημαντικό η συνθήκη πλαίσιο να εφαρμοστεί ακριβώς όπως έχει προβλεφθεί και να συμφωνούμε απολύτως, τα δύο θεσμικά όργανα δηλαδή, στην ερμηνεία της. Επ' αυτού ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας. Η συνθήκη αποδίδει σημασία στις διαθεσμικές συμφωνίες. Πρέπει να είμαστε λοιπόν σε επαγρύπνηση και από πλευράς, όπως είπα, της Κομισιόν θεωρούμε την συμφωνία αυτή ως εξαιρετική. Ένα συνάδελφο είχε ζητήσει να λάβει το λόγο. Ε, Δυστυχώ αντέστρεψα λίγο την σειρά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ξέρω κατά πόσο μπορούμε να βρούμε μια ισορροπία. Γιατί εγώ καταλαβαίνω το επιχείρημα του κύριου Νταφ και την τροπολογία, της, την τροπολογία του που λέει ότι ενισχύεται ο ρόλος στην εξωτερική πολιτική αλλά μετά λέει με εξαίρεση τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση στην διατύπωση του κειμένου. Συγχρόνως, ο κύριος Αγγέλη και ο κύριος Ρομέρο μας λένε ότι είναι ένα κείμενο στο οποίο καταλήξαμε μετά από λεπτές ε, ισορροπίες. Οπότε, καταλαβαίνω το επιχείρημα που λέω ότι δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε μια συμφωνία η οποία επιτεύχθη με τόσο μεγάλη προσπάθεια από όλες τις πολιτικές ομάδες όπου προσπαθήσαμε να βρούμε λύσεις Εγώ πιστεύω ότι μόνο σε πνεύμα συνένεσης μπορούμε να ψηφίσουμε. Οπότε ζητάω από τον κύριο Ραγγέλ και τον κύριο Νταφ. Μήπως η τροπολογία του κύριου Νταφ θα μπορούσε να σωθεί ως εξής. εκεί που λέει και ενισχύει το ρόλο του στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τελεία, να προσθέσουμε με τις ρυθμιστικές διευκρινήσεις που αντιστοιχούν στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Ρυθμιστικές διευκρινήσεις που υπάρχουν ήδη. Για να μην υπάρχει αντίφαση ανάμεσα μέσα στο κείμενο. Αντί δηλαδή να βγάλουμε όλη την ε, τελευταία παράγραφο, τις τρει τελευταίες γραμμές, να πούμε ότι ενισχύει το ρόλο του στην εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τις ρυθμιστικέ διευκρινήσει που αντιστοιχούν στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Έτσι διευκολύνεται νομίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι σώζεται και το πνεύμα το οποίο επιθυμεί να δει ο κύριος Ντάφ. Εσείς κύριε Ντάφ θέλετε να λάβετε το λόγο. Κοιτάξτε. Ναι. Θα προτιμούσα να πω ο ρόλος του σε ορισμένες εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης περιλαμβανομένης της ΚΕΠΑ, της κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Αν όμως ο κύριος Ραγγέλ υποβάλει κάποια ευφιέστερη πρόταση ε, να την εξετάσω. Εσείς κύριε Αντζέλη. Δύο σχόλια. Θα έρθω στα όσα είπε ο νομίζω ότι μπορούμε να αντιδεχτούμε την πρόταση αυτή που σέβεται το κείμενο. Και την έννοια του τι είναι κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Νομίζω ότι <clears throat> κάτι μέσα στα πλαίσια αυτής της φόρμουλας, δεν ξέρω βέβαια πώς θα το πω στα αγγλικά, αλλά κάτι ε, με την έννοια αυτή. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει δεκτό. αφού ενισχύει την ιδέα ότι η κοινή εξωτερική πολιτική και ασφάλειας είναι διαφορετικό, κάτι διαφορετικό από τις εξωτερικές σχέσεις συνολικά. Νομίζω ότι αυτό αρκεί. Να αντικαταστήσουμε δηλαδή μια έκφραση που περιλαμβάνει μια εξαίρεση με μια έκφραση πιο ουδέτερη. Ας πούμε περιλαμβανομένης της κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Μου φαίνεται κάπως πιο ευρωπαϊκή διατύπωση αυτή. Ναι, ναι, ε, και, ε, και εγώ την δέχομαι αυτή την πρόταση. Μη Eh, Σαν να διαγράφεται μια συνένεση των πολιτικών ομάδων. Αλλά για ποια τροπολογία μιλούμε. Την ένα. Ah, Καλώς λοιπόν. Ναι, εσείς. Για τη μας ξανά την διατύπωση αυτή. Επαναλάβετε τη, τη διατύπωση αυτή. Ναι, ναι, παρακαλώ κύριε Αντζέλ. Δεν θυμάμαι ακριβώς την κάθε λέξη, αλλά έλεγε περίπου περιλαμβανομένης έλεγε της ΚΕΠΑ περιλαμβανομένης της κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας σύμφωνα με ναι τις οικίες διατάξεις είχε πει προηγουμένως ο, ο εισηγητής. Μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Ας αρχίσουμε λοιπόν τότε. Κείμενο προσαρμογή του κανονισμού στη Συμφωνία Πλαίσιο στις σχέσεις Κοινοβουλίου Κομισιών. Τροπολογία 14. Αφορά το άρθρο 9, παράγραφος 2 υπέρ. κατά αποχές με μία ψήφο κατά αποσύρεται η παραθμόν 1 15 του εισηγητή 23 υπέρ κατά αποχές με ψήφο κατά εγκρίνεται η δύο αποσύρθηκε Τροπολογία 3, άρθρο 35. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται ομόφωνα. Τροπολογία 4 του εισηγητή. Άρθρο 43. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16 του εισηγητή. Άρθρο 44. Υπέρ κατά ένας. Εγκρίνεται η 5 σύρθηκε. 6. Άρθρο 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 17 και 19. Υπέρ κατά μία πιο κατά αποχές εγκρίνεται. Η 18 καταπίπτει, η 8 αποσύρθηκε, Τροπολογία 20. Υπέρ κατά αποχές. Με μία αποχή εγκρίθηκε. Αποσύρθηκε η εννέα. 10. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 12 αποσύρθηκε 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 αποσύρθηκε 22 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται 23 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ομόφωνα. Το χειροκρότημα στο τέλος. Θα ψήσουμε την προσαρμογή του κανονισμού στον αναφερμένο κείμενο. η αναθεώρηση του Συμφωνίας Πλαίσιο για τη σχέση Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιτροπής τέσσερις τροπολογίες. Πρώτη είναι του συναδέλφου Νταφ. Υπέρ. Νταφ. Ε, είπα η πρώτη είναι η τροπολογία 2. Η τροπολογία 2 του συναδέλφου Νταφ στην παράγραφο 3, 4, 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3. υπέρ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. τέσσερα Νταφ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τροπολογία υπάρχει μόνο ένα με την προφορική τροπολογία υπέρ κατά ένας αποχές εγκρίνεται τελική ψήφος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τώρα πρέπει να χειροκροτήσουμε τη Σανφό Ραγκέρα για την πολύ καλή δουλειά του και στις διαπραγματεύσεις έχουμε να ψηφίσουμε Είμαστε στο 8. Διορθωτικό προπολογισμό, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο Τμήμα 3 Επιτροπή, Τμήμα 10 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Η Επιτροπή μα θα γνωμοδοτήσει προ την Επιτροπή Προπολογισμών για τον διορθωτικό προπολογισμό 6-2010 και της Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Μπορούμε να υποβάλουμε και τροπολογίες. Υποβάλαμε τροπολογίες Ο Σάνφος Βέροφστατ δεν είναι παρόν. Τυπικά δεν ορίσαμε εισηγητή τον κύριο Βέροφστατ, αλλά de facto αυτός μας εκπροσώπησε. που μπορούμε και επίσημα να ορίσουμε τον κύριο Βεροστά τον συζητητή αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Απουσία του κύριου Βεροστάτ Ερχόμαστε στη συζήτηση. Πρώτο συνάδελφο Νταφ. Πρόεδρε. Ο κύριο Βεροστάτ ευχαριστεί την Επιτροπή που τον όρισε. Ζητώ συγγνώμη γιατί δεν μπορεί να είναι παρόν σήμερα. εγγυάται ότι οι τροπολογίες που προτείνει συμφωνούν είναι ακριβώς οι ίδιες Μέσα Με τις τροπολογίες του κύριου Μπροκ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων υπάρχει λοιπόν διακομματική συνένεση και ελπίζω να είναι δυνατόν να ψηφιστούν ένα μπλοκ και να εγκριθούν. Πρόεδρος. Μπορούμε να ψηφίσουμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Νταφ. Οι τροπολογίες είναι 7. Συμφωνημένες με τις ομάδες. Πιστεύω, αν δεν υπάρχει αντίθεση, ότι πρέπει να ψηφίσουμε ένα μπλοκ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. μία ψήφο κατά εγκρίνεται. Τελική ψήφος στη γνωμοδότηση. Υπέρ. Κατά. Ένας κατά αποχές. Εγκρίθηκε. Τελείωσε η σημερινή μας συνεδρίαση. Παρακαλώ να μείνουν οι συντονιστές. Σας θυμίζω ότι σήμερα σε αυτή την αίθουσα ήρθαμε επειδή είχαμε καλέσει και άλλα άτομα. Αύριο θα είμαστε σε άλλη αίθουσα. Αυτό η Γραμματεία και εγώ σας παρακαλούμε να μην αφήσετε τίποτε εδώ γιατί δεν θα είστε το πρωί εδώ. Επαναλαμβάνω θα είμαστε σε άλλη αίθουσα αύριο. Πέρα στις συνεδρίες.